So, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα. Πρώτο θέμα, το σημείο παριθμών 8. Έχουμε συζήτηση με τη Φιλανδική Προεδρία και χαίρομαι πολύ που έχουμε εδώ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου της ε, Φιλανδίας, τον κύριο Σκινάρη ο οποίος είναι εδώ μαζί μου για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας και να συζητήσει μαζί μας. Αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις στον τομέα του εμπορίου. Εχθές ε, συζητήσαμε λίγο κάποιες εξ αυτών, το θέμα του Μερκοσούρ και νομίζω ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία για το επόμενο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει πολλή συζήτηση φυσικά και θα έχουμε και την κύρωση της συμφωνίας ε, του Βιετνάμ και ελπίζω να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εργασίες και από αυτού σύντομα. Δυστυχώς υπάρχει και το Brexit και θα πρέπει να συζητήσουμε και ε, τη συμφωνία εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά Υπάρχει επίσης και το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, ε, όπου υπάρχει κάποια σύγχυση τα τελευταία χρόνια και κάποιος εκνευρισμός όσον αφορά τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον ΠΟΕ. Και έχουμε επίσης και ένα σημαντικό νομοθέτημα για τα νέα μέλη. Ε, εγκρίναμε πριν από δύο χρόνια το κανονισμό για τους ελέγχους ε, προϊόντων ε, διπλής ε, χρήσης και τις εξαγωγές τους και θέλουμε να έχουμε και πληροφορίες, πληροφορική και τεχνολογία, να συμπεριλάβουμε και το hardware και το software στο σύστημα των ελέγχων, ώστε οι περιορισμοί που είδαμε στην Αραβική Άνοιξη μέσω της ευρωπαϊκής τεχνολογίας για την αντιπολίτευση να μην ε, επαναληφθούν στο μέλλον. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κοινή θέση για δύο χρόνια. Τώρα υπάρχει κοινή θέση και ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθεσία αυτή στη διάρκεια τη Φιλανδική Προεδρία. Πολλά πράγματα λοιπόν, πολλά καθήκοντα και φυσικά ε, ο χρόνος της Φιλανδικής Προεδρίας είναι πολύ περιορισμένος και προσβλέπουμε φυσικά στη συνεργασία μαζί σα για αυτά τα θέματα. Να δώσω τώρα το λόγο σε εσά για να μας κάνετε την παρουσίασή σας για τις ε, απόψει σας και τις ιδέε σα. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάγκε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι προφανώς τιμή και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να συζητώ μαζί σας και να σας παρουσιάσω το θεματολόγιο της Φιλανδίας και φυσικά να ανταλλάξουμε απόψεις και σκέψεις για την εμπορική πολιτική εν γέννη. Όπως ε, ακούστηκε, το εξωτερικό εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινότητας Είμαστε το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ του κόσμου και ο μεγαλύτερος ε, παρασκευαστής ε, ε, εμπορευμάτων αλλά και πάροχος υπηρεσιών. Είμαστε και ο μεγαλύτερος επενδυτής και ο μεγαλύτερος παραλήπτης ξένων επενδύσεων. Είμαστε ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός εταίρος για πάνω από 80 χώρες. Και οι πραγματικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και πρωτοβουλίε όπως τα πάντα εκτός από όπλα δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές υποστηρίζουν 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Περίπου 14 εκατομμύρια από αυτούς τους εργαζομένους είναι γυναίκες. Μία στις 7 θέσεις εργασίας εξαρτάται από τις εξαγωγές. Αυτές οι εξαγωγές υποστηρίζουν επίσης 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεριλαμβάνουν φυσικά και αναπτυσσόμενες χώρες. Το εμπόριο είναι μία πρόταση win-win. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, οδηγεί στην ανάπτυξη και βελτιώνει το βιωτικό επίπεδο. Μειώνει την ένδια και φυσικά ενισχύει τον ανταγωνισμό. Ενώνει ανθρώπους. Επίσης προωθεί τις καινοτομίες και βοηθά την ενίσχυση. τα αποτελέσματα τα οποία ε, είναι αμοιβαία επωφελή ε, οδηγούν σε διαρκή αποτελέσματα, διαρκή ωφέλη και πραγματικά το ε, να σκεφτόμαστε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει είναι λανθασμένος τρόπος, λανθασμένη οπτική για το εμπόριο. Επίσης πρέπει να προωθούμε και τις ευρωπαϊκές αξίες. Το εμπόριο πρέπει να αντανακλά τις δεσμεύσεις μας για ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει επίσης να διατηρεί τα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικών και καταναλωτικών ε, θεμάτων και προστασίας. Και σήμερα η νομιμοποίηση της εμπορικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέει από την ε, λαϊκή υποστήριξη των εμπόρων και των πολιτών και των επιχειρήσεων η Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ε, συζήτηση πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της διαδικασίας λήψη αποφάσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ευρία συνένεση για το θεματολόγιο του εμπορίου. Αυτό μα προσφέρει ε, ισχυρά θεμέλια για να ενισχύσουμε τα συμφέροντά μας στον κόσμο. Προσβλέπω φυσικά στη συζήτησή μας σήμερα και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά τους επόμενους μήνες ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών μας αξιών. Τις αξίες ε, τις ανέφερα ήδη, αλλά είναι ιδιαίτερα παρούσες ε, στο πρόγραμμα της κυβέρνησής μας, το οποίο ισχύει από τον Ιούνιο. Το πρόγραμμα επισημαίνει τη βιωσιμότητα και την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη. Πιστεύω ότι όλοι ε, συμμεριζόμαστε αυτούς τους στόχους. Επισημαίνουμε τη σημασία ενός εμπορίου που θα είναι φιλόδοξο, ανοιχτό και θα βασίζεται σε κανόνες και θα έχουμε και κατάλληλη πολιτική επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καιρό ε, παγκοσμίων εντάσεων και αυξανόμενο προστατευτισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπίζεται το σύστημα πολυμερούς εμπορίου και τους κοινού κανόνες, καθώς επίσης και να παραμείνει ανοιχτή ε, στο διεθνές εμπόριο. Ο ΠΟΕ είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ε, παγκόσμιας διακυβέρνησης και πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί. Δεσμευόμαστε λοιπόν για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει μια σειρά από προτάσεις και αυτή τη στιγμή το πιο πιαστικό θέμα αφορά την επίλυση διαφορών και τον ε, αντίστοιχο φόρεα, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι φαίνεται ότι αυτός ο φορέας ε, για την άσκηση εφέσεων ε, δεν θα προχωρήσει. Ε, το σύστημα του εμπορίου λειτουργούσε εδώ και πάνω από 40 χρόνια ε, με, χωρίς δεσμευτική ε, λύση για επίλυση διαφορών αλλά οι χώρες ε, πλέον δεσμεύτηκαν ε, να ανοίξουν και να απελευθερώσουν το εμπόριο. Αυτές ε, δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλες προϋποθέσεις. Επομένως πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάποιες προτάσεις, έκανε μάλλον τις προτάσεις και θα δούμε τους επόμενους μήνες εάν θα υποστηριχθούν και από τα υπόλοιπα μέλη. Είναι σαφές κατά την άποψή μου ότι σε μια κατάσταση όπου τα μέλη αρχίζουν να ε, αγνοούν τους κανόνες του ΠΟΕ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, οι μικροί και πιο ευάλωτοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πληγούν περισσότερο. Οι σχέσεις μας εμπορίου και επενδύσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, παραδοσιακά ήταν πολύ μεγάλε και αμοιβαία επωφελεί. Οι οικονομίε μα ε, συνδέονται άμεσα η Διατλαντική Συμμαχία ήταν ε, η ραχοκοκαλιά της διεθνούς ασφάλειας και του διεθνούς συστήματος. Παρά τις παρούσες δυσκολίες ε, στις σχέσεις μας, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη ε, σχέσεις μας ε, για να προχωρήσουμε το θεματολόγιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παρούσες εντέσεις ε, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτείων είναι γνωστές. δασμοί στο χάλιβα και στο, αλουμούλιο, στο αλουμίνιο και επιβάλλονται από μια αμφίσιμη ερμηνεία της εθνικής ασφάλειας. Τα μέτρα που αφορούν εισαγωγές ευρωπαϊκών οχημάτων και ανταλλακτικών εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα, είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε επί τη βάση μιας ισορροπημένης επικοδομητικής σχέσης μεταξύ ίσων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για βιομηχανικούς δασμούς και αξιολόγηση της συμμόρφωσης βάσει της εντολής του Συμβουλίου. Επίσης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε σε διεθνές επίπεδο, αναζητώντας λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, ε, προς τρίτες χώρες. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, με τον ίδιο ε, τρόπο με τον οποίο το κάναμε και στο παρελθόν, συμβατό προς τον ΠΟΕ. Να περάσω τώρα στην Κίνα. Η Κίνα είναι και πολύ σημαντικός εταίρος που παρήχει τεράστιες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ε, παγκόσμια δύναμη η οποία ε, δημιουργεί και πολλές προκλήσεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις εμπορικές πρακτικές της Κίνας. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην πρόσβαση στις αγορές. Υπάρχει κρατική παρέμβαση η οποία δημιουργεί στρεβλώσεις, ε, υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας ε, και παραβιάσεις ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Αντί λοιπόν να προχωρούν στο δρόμο του ανοίγματο, υψώνουν νέους φραγμούς. Είναι επίσης σαφές ότι η Κίνα, όπως και οποιοδήποτε άλλος, πρέπει να τηρεί τους κανόνες. Προσπαθούμε να βρούμε πολυμερείς λύσεις, ελπίζουμε μαζί με την Κίνα. Ωστόσο, ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτούμε και ευρωπαϊκές λύσεις. Να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία για να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να επιτύχουμε και στην Κίνα αλλά και οπουδήποτε αλλού. Μας ενδιαφέρει και διεσμευόμαστε φυσικά ε, για τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Συμφωνιών στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις εν εξελίξη, όπως για παράδειγμα με τη Χιλή, το Μεξικό, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ινδονησία. Ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι η πρόσφατη ε, υπογραφή της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου και της ε, Συμφωνίας Προστασίας των Επενδύσεων με το Βιετνάμ. Η συμφωνία ενισχύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας του σαφού οικονομικού ωφέλου. Οι συμφωνίε αυτές ε, έχουν στόχο να ενισχύσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος ε, και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η δέσμευση του Βιετνάμ στη διαδικασία μέχρι τώρα είναι ε, ευπρόσδεκτη φυσικά. Η πρόσφατη κύρωση της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις είναι εξαιρετικό παράδειγμα ε, του πώς οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα πρότυπα. Εάν το Συμβούλιο συνενέσει σε αυτές τις συμφωνίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε κατάλληλα εργαλεία για να προωθήσουμε τις αξίες μας και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που ξέρω ότι έχουν πολλοί από εσά όσον αφορά τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα εργασίας στο Βιετνάμ. Οι συμφωνίες αυτές έχουν ήδη καταδείξει ότι ε, παρέχουν μόχλευση και χωρίς αυτές η μόχλευση αυτή ε, χάνεται. Η πολιτική συμφωνία με τη Μερκοσούρ, με τις χώρες του Μερκοσούρ είναι ε, πάρα πολύ σημαντική και από πολλές απόψεις θεωρείται ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όχι μόνο από οικονομική σκοπιά, αλλά και από πολιτική σκοπιά. Ήταν ε, στρατηγικός ρόλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για πάνω από 20 χρόνια. Στέλνει ένα μήνυμα ότι σε καιρού αυξανόμενου παγκόσμιου προστατευτισμού υπάρχουν χώρε οι οποίε είναι διατεθειμένε να δεσμευτούν και να ανοίξουν το εμπόριο αντί να κλείσουν τι αγορέ του. Όσον αφορά τη συμφωνία, πρέπει ακόμα να δούμε τα κείμενα τα οποία έτυχαν διαπραγμάτευσης για να αξιολογήσουμε κατάλληλα τον αντίκτυπό τους. Αυτό περιλαμβάνει ε, και την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ωστόσο, η συμφωνία θα ανοίξει πολύ σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες ε, του Μερκοσούρ. Πέραν του εμπορίου, η μελλοντική συμφωνία θα παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για πολιτικό διάλογο και συνεργασία και στενότερη δέσμευση σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει και την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η Βραζιλία και άλλες χώρες του Μερκοσούρ δεσμεύονται μέσω της συμφωνίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Το ξέρω ότι αυτό είναι βασικό θέμα για το Κοινοβούλιο και για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Δεδομένων και των πυρκαγιών ε, οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή μένονται στον Αμαζόνιο, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως ε, αυτή με το Μερκοσούρ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι χώρες όπως η Βραζιλία θα σέβονται τις διεθνείς τους δεσμεύσεις. Γενικότερα τώρα πρέπει να προωθήσουμε την ολοκλήρωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην ε, ε, παγκόσμια οικονομία. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την Αφρική, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης εντός της Αφρικής. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η περιοχή ελευθέρου εμπορίου της Αφρικανικής Υπήρου ε, κερδίζει αυτή τη στιγμή εντυπωσιακή όθηση. Όσον αφορά το εμπόριο λοιπόν, ε, συμβαίνουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα είναι εξίσου σημαντικό να εστιάσουμε περισσότερο στην κατάλληλη εφαρμογή ε, και υλοποίηση των κείμενων συμφωνιών. Συνεπώς, θέλουμε να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη των εμπορικών συμφωνιών θα χρησιμοποιούνται πλήρως από τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας θα εφαρμόζουν τους κανόνες και θα σέβονται τις δεσμεύσεις ε, που ε, συμφώνησαν να σεβαστούν. Με βάση τη συνολικότερη έμφαση προς τη βιωσιμότητα, πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, την ισότητα του φύλου και τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μόνο μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τους εταίρους μας. Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουμε και τις εργασίες ε, του κεφαλαίου εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές συμφωνίες ε, μέσω ανάπτυξης ε, ενός μηχανισμού προσφυγών που θα είναι πιο εξορθολογισμένους, για παράδειγμα. αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι η εφαρμογή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σχέση μας με το Μερκοσούρ. Είναι πολύ καλό να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ήδη καταλήξει σε θετικές δεσμεύσεις από πλευράς Βιετνάμ. Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμες αλυσίδες αξιών είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τη Φιλανδία. Σκοπεύουμε να οργανώσουμε μια διάσκεψη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο με στόχο να προχωρήσουμε τη συζήτηση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η καταπολέμηση και ο μετριασμός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι ε, μια ισχυρή ε, κυρίαρχη προτεραιότητα για τη Φιλανδική Προεδρία. Σε όλες μας τις εμπορικές συμφωνίες και στις κείμενες αλλά και σε αυτές οι οποίες είναι υπό διαπραγμάτευση δεσμευόμαστε για τη Συμφωνία του Παρισιού και τη συνεργασία σε θέματα κλίματος. Ήγηκε λοιπόν η ώρα να προχωρήσουμε προς την εφαρμογή. Υπάρχουν ευκαιρίες ε, για την απελευθέρωση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και ε, την προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα. Είναι επίσης επιτακτική σημασία ε, να προχωρήσει το θέμα της τιμολόγησης του άνθρακα παγκοσμίω και να προχωρήσουμε και με τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων. Αντί για περιορισμό του εμπορίου με μέτρα στα σύνορα, θέλουμε να ανοίξουμε περαιτέρω της αγοράς για να υπάρχουν ε, εισαγωγή και εξαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών παγκοσμίω. Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο Κοινοβούλιο οι συνάδελφοι υπουργοί μίλησαν νωρίτερα για την ανάγκη να αναπτύξουμε περαιτέρω την ενιαία αγορά. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τις υπηρεσίες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα έχουν αντίκτυπο φυσικά και στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοίχως, η παρούσα και μελλοντική εμπορική νομοθεσία θα πρέπει να ε, σχεδιαστεί έχοντας κατά νου την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία να ε, δείξει ηγετικό ρόλο και ευθύνη για να ανοίξει το δρόμο για το βιώσιμο μέλλον. Αυτό ε, σημαίνει ότι πέραν ε, του κοινού οράματος ε, πρέπει να υπάρξουν κοινέ προσπάθειες, κοινέ δράσεις και πιο σημαντικό από όλα κοινή εφαρμογή η οποία θα έχει συμφωνηθεί από κοινού. Για άλλη μια φορά προσβλέπω στις συζητήσεις μας σήμερα και στην περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για αυτή την εκτεταμένη και εξαντλητική επισκόπηση για τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας σας το επόμενο διάστημα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αρχίζουμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ε, ομάδων, τους συντονιστές, ε, δύο λεπτά. Ε, θα έχετε την ευκαιρία μετά να απαντήσετε και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά ο συντονιστής, ο κύριος Κριστόφ Χάνζεν. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε Λάγκε. Ευχαριστώ και σας Υπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Έχω Πολύ σύντομε ερωτήσει και λίγε. Πρώτον, η Φιλανδική Προεδρία προτίθεται να προχωρήσει ε, στη ε, συμφωνία με την Ταϊβάν. Πρώτη ερώτηση. Και για τα είδη χρήση, χρήσης ε, η Φιλανδική Προεδρία προτίθεται να κλείσει το φάκελο αυτό. Θα δείξει την απαραίτητη ευελιξία το Συμβούλιο για να γίνει. Και η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με τα ε, όσα μάθατε από τα κράτη-μέλη που βολιδοσκοπήσατε το ε, καλοκαίρι, τι ε, θα κάνετε για τις διεθνείς προμήθειες και το αντίστοιχο μέσο. Από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ. Σας χαίρω για την νέα σας φιλανδική κυβέρνηση με το τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. Δύο πράγματα θέλω να θίξω. Προφανώς το πρώτο είναι το Mercosur που ε, ε, μας απασχολεί πάρα πολύ και μας ανησυχεί και το Κοινοβούλιο και την πολιτική μου ομάδα. Μετά τις ενές διακοπές ε, τα ακούσαμε όλα αυτά να απασχολούν την κοινή γνώμη σε όλες μας τις εκλογικές περιφέρειες. Και υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιδράσεις. Η πρώτη λέει ότι θα πρέπει να τρέξουμε το Μερκοσούρ γιατί έτσι θα σταματήσουμε τις δασικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Και η άλλη αντίδραση λέει το αντίθετο. Όχι, να μην κυρώσουμε τη συμφωνία Μερκοσούρ, να τη σταματήσουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει κανένα από τα δύο αυτά. Δεν βλέπω καμία απόδειξη ότι αν είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα θα σταματούσαμε τις πυρκαγιές. Αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στρατηγικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Συμφωνία Μερκοσούρ πριν την κυρώσουμε, έτσι ώστε ουσιαστικά να εφαρμόσει τη Συμφωνία των Παρισίων ε, και ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών κτλ. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις ε, πριν από την κύρωση. Και ρωτώ τη Φιλανδική Προεδρία. Εσείς είστε διατεθειμένοι να αρχίσετε αυτή την πολιτική συζήτηση και στο Συμβούλιο. Δεύτερη ε, ερώτηση, γενικά ε, για την κλιματική πολιτική. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξη η κυβέρνησή σας ε, για να έχουμε ουδέτερο το κλίμα και την πολιτική μέχρι το 2035. Εδώ έχουμε πλειοψηφία για το 2050. Τι σημαίνει αυτό, κλιματικό νόμο, νομοθεσία, περισσότερες φιλοδοξίες για το 2050 και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το σύστημα εμπορία εκπομπών, στο ETS, και σε ό,τι αφορά και τη διαρροή λεγόμενη άφακα που φεύγουν ε, οι ε, πολλοί ρηπογόνε ε, επιχειρήσεις και βιομηχανίε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υψηλού στόχου στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύουμε και τη βιομηχανία μα Και στο Κοινοβούλιο τούτου δύο επιτροπή θα πρέπει να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια, ε, όπως και εσεί, στο Συμβούλιο είστε πρόθυμοι να το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κάλσπο από την ομάδα Renew Europe. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και μας εμπνέει πάρα πολύ το να σας ακούμε. Ακούμε το φιλανδικό παράδειγμα, πώς καταφέρατε εσείς στη χώρα σας να συνδυάσετε το εμπόριο και την αναπτυξιακή πολιτική ως στρατηγική για μια παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και είμαι βεβαία ότι αυτό θα μας εμπνεύσει και μας ε, στη δουλειά μας εδώ στην καθημερινή μας εργασία στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Θα σας παρακαλούσα να εμβαθύνετε λίγο προς το χρονοδιάγραμμα. Πώς το βλέπετε αυτό το φθινόπωρο. Ποια είναι τα σχέδιά σας ε, χρονικά για να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους επόμενους μήνες. Και επίσης θα ήθελα να πω δύο λόγια αυτό που συζητούμε και μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες και θα κυριαρχήσει και τον επόμενο μήνα, γι' αυτό είναι όντως το θέμα του Μερκοσούρ και της κλιματικής αλλαγής από τη μια και του εμπορίου από την άλλη. Εμείς πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο τι παραμονές της υπογραφής μια συμφωνίας, αλλά και μετά την υπογραφή της. Αυτή είναι μία από τις ε, βασικές συζητήσει που θα γίνει στην κοινή γνώμη, πιστεύω, και μεταξύ των πολιτικών και μεταξύ των πολιτών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν δεν γίνει αυτή η συζήτηση σωστά, ο κόσμος δεν θα καταλάβει ότι είναι σημαντικό το εμπόριο και μπορεί να βοηθήσει, όπως πιστεύουμε εμείς. Ευχαριστώ. a lot. Ευχαριστώ πολύ από τους Πρασίνους η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλωσορίσατε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, βλέπουμε να αλλάζει λίγο το ύφος των όσων λέτε και, το, το περιεχόμενο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό που ε, ε, οι ασχολούμενοι με το εμπόριο υποστήριζαν ότι το εμπόριο είναι εμπόριο και όλα τα υπόλοιπα είναι άλλων θέματα. Τώρα έχουμε όμως το 2030 το θεματολόγιο, θα πρέπει να συνδέσουμε περισσότερο ακόμα το εμπόριο με την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο με τη γεωργία, το εμπόριο με άλλα θέματα, με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό όμως και να είναι αμοιβαία επωφελή ε, όλα αυτά και το ελεύθερο εμπόριο, πρέπει να δράσουμε. Και εμείς ως Φιλανδοί αυτό το υποστηρίζουμε και ούτε η Σουηδία θα ήταν αυτό που είναι σήμερα αν δεν είχαμε ανοίξει το εμπόριο Εμεί στην αρχή του 20ου αιώνα. Τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Για να παραμείνουν αυτό όμως αμοιβαίως υποφελή θα πρέπει η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι ενταγμένη στις εμπορικές πολιτικές. Υπάρχουν κάποια θέματα επίκαιρα που ανάφεραν οι συνάδελφοι. Κοιτώ τώρα τη συμφωνία Μερκοσούρ Το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, επανειλημμένα ε, αναφέρει τον όρο «shall». The parties shall, δηλαδή εσείς που είστε και νομικός, πώς το εξηγείτε αυτό, ποιες είναι οι υποχρεώσεις των διαφόρων μερών. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στην εφαρμογή όλων αυτών που οφείλουν να κάνουν τα κράτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, για να σημαίνει κάτι αυτό και να μπορεί να επιβάλλεται στην πράξη. Γιατί σε αυτό το κείμενο για το συγκεκριμένο κεφάλαιο που είναι 50 σελίδες, δεν βλέπω καμία επιβολή. Παρόλη την γλωσσική αυτή διατύπωση ότι τα κράτη ή τα μέρη οφείλουν, οφείλουν πώς θα το επιβάλλουμε. για να μην επιδερωθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη χρήση γης, τις δασικές πυρκαγιές, την αποψήλωση των δασών και την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών. Ε, ο κύριος Βέλης από την ομάδα ID. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Φιλανδό Υπουργό για την εξαιρετική του ομιλία. Ε, θα ήθελα να πω το εξή. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν καλός φίλος και πελάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο εμπόριο των αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία είχαμε πλεόνασμα 44 δισεκατομμύρια στερλίνες κάθε χρόνο ε, ε, στη δεκαετία μέχρι το 2017. Τα τελευταία 10 χρόνια Ε, ε, η Ευρώπη είχε 489 δισεκατομμύρια ε, πλεόνασμα. Εμείς έχουμε δώσει δισεκατομμύρια και στον κοινοτικό προϋπολογισμό τα τελευταία 10 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο ως καθαρός συνεισφορέας έδωσε περίπου 90 δισεκατομμύρια στερλίνες. Μετά την επιστροφή των χρημάτων, έχουν αφαιρεθεί αυτά που παίρνουμε πίσω. Είναι μία από τις έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σέβεται το όρο του ΝΑΤΟ για 2% στρατιωτικών δαπανών. Ε, η συμφωνία για το Brexit θεωρείται χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών από ε, ε, την κοινή μας γνώμη και το backstop και ε, ο λογαριασμός που μας έχετε βγάλει σε δισεκατομμύρια ως προϋπόθεση για να συζητήσουμε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και επίσης θέλει να συνδέσει τις Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στα στρατιωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε και η κυρία Βαντρελάιν η ίδια ότι ε, θα συμμετέχουν στον Ευρωστρατό. Και ε, πού είναι η νομοθεσία και οι κανόνες ε, που θα μας επιβάλλεται. Δεν θα μπορεί ο Βρετανικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον του. Ερωτώ λοιπόν τον Φιλανδό Υπουργό και τον κύριο Γιούνκερ και την κυρία Φόντερ Λάιν το άρθρο 24 του ΓΚΑΤ, μήπως το έχετε σκεφτεί για να λυθεί το θέμα των ελλαδικών συνόρων, για να προχωρήσουμε ε, καλή πίστη σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Βρετανικό λαό. Και αν όχι, γιατί όχι. Έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Ε, ήσασταν μία εγγεγραμμένος εσείς από την ID. Είναι ο κύριος Κόφουτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την ομιλία σας. Δύο ερωτήσεις έχω μόνο. Ερώτηση πρώτη. Όταν συζητούμε τις εμπορικές συμφωνίες, συχνά είναι ε, είτε το εμπόριο μόνο του, είτε και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Και τα δύο είναι σημαντικά όμως, όχι μόνο το εμπόριο. Και φυσικά και οι εργαζόμενοι και το κλίμα. Εσείς όλα αυτά πώς το βλέπετε αυτό το δίλημα ενώ και πώς το χειρίζεστε. Ε, πρόσφατα αναφερθήκατε και στην ομιλία σας σύντομα, θέλω λίγο να επεκταθείτε. Μιλήσατε και για την Αφρική πάρα πολύ σύντομα στην ομιλία σας και εκεί θα ήθελα λίγο να επεκταθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από το ECR ο κύριος Χέρτ Πουρζουά. Ευχαριστώ Υπουργέ. Συμφωνώ με τις βασικές προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας και έχω και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτο, για το Brexit. Έχετε σχέδια για να προετοιμάσετε τις μελλοντικές σχέσεις αν υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία. Θα πρέπει να εξάγουμε με βάση τους κανένας των του ΠΟΕ με τεράστιους δασμούς εισαγωγικούς. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρξει το λεγόμενο σκληρό Brexit θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι οι μελλοντικέ μας σχέσεις και τουλάχιστον μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών πρέπει να υπάρχει. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν σχέδια να συνεχιστεί ο διάλογος με τον Πρόεδρο σε επίπεδο Πρόεδρων, δηλαδή Πρόεδρου Ιούνκερ με τον Πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει μια ιδέα να ε, συνεχίσουμε μια περιορισμένη συμφωνία για τα βιομηχανικά αγαθά και κατά τα άλλα να έχουμε σκληρή στάση για τα αντίπεινα. Αλλά έχει έρθει η ώρα να αρχίσει ο διάλογος, νομίζω. Ε, μας συμφέρει και τους δύο. Για την Κίνα. να ε, αντιδράσουμε κατά το dumping στις τιμές, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε και συμφωνία επενδυτική που να βασίζεται σε αμοιβαιότητα. Τώρα οι εταιρείε μα ε, μεταφέρουν τεχνογνωσία και τεχνολογία όταν πηγαίνουν στην Κίνα. Ενώ όταν έρχονται εδώ οι Κινέζοι δεν υπάρχει καμία αμοιβαιότητα. Πολύ μεγάλη ε, ε, σημασία και αυτό. Και τέλος για την Ινδία. Από το 2013 έχει σταματήσει ο διάλογος για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Σχεδιάζεται να έρθει σε επαφή με την Ινδική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουτ Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της ε, ε, εμπορικής πολιτικής, έτσι όπως τη βλέπει η Φιλανδική Προεδρία. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το σύστημα βασισμένο σε κανόνες. Πρέπει να είναι πραγματικά βασισμένο σε αληθινούς κανόνες. Είμαι από μια χώρα όπου κάποτε επικρατούσε το σκεπτικό ότι οι κανόνες είναι για πάντα. Και οι κανόνες βέβαια και οι προσδοκίες των ανθρώπων αλλάζουν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό, αυτή την πεποίθηση όπως άλλαξε στη χώρα μου έτσι ελπίζω να αλλάξει και εδώ. Οι παγκόσμιες αλυσίδες αξιών είναι προϋποθέσεις οι οποίες δεν είχαν την ε, ύψιστη προτεραιότητα στον ΠΟΕ μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πώς η Φιλανδική Προεδρία και γενικότερα το Συμβούλιο σκοπεύει να προχωρήσει έτσι ώστε να αποκτήσουμε κοινούς κανόνες να υπενθυμίσω ότι φυσικά η Κίνα και η Ινδία έχουν διαφορετική προσέγγιση σε αυτούς τους κανόνες που δημιουργήθηκαν 20-30 χρόνια πριν. Δεν θεωρείτε πως ε, έχουμε όλοι ευθύνη για επικαιροποίηση των ε, κανόνων του ΠΟΕ. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο το έργο, είναι μεγάλη πρόκληση. καθώς επίσης και το πώς θα προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Έπειτα, πώς θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο την εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, με ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τις πτυχές της νέας νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έχετε έξι λεπτά να απαντήσετε στον πρώτο κύκλο ερωτήσεων, γιατί έχουν ζητήσει άλλοι 11 συνάδελφοι το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πολλές από τις ερωτήσεις ε, τις ε, άγγιξα στην παρουσίασή μου, θα προσπαθήσω όμως να καλύψω όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές. Ε, καταρχάς, ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα βασισμένο σε κανόνες και τις ε, αξίες που πρεσβεύουμε. Η κυβέρνηση της Φιλανδίας πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε αξίες. Αυτό αφορά και την εμπορική πολιτική. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ μια εμπορική συμφωνία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη ε, τις περιβαλλοντικέ επιτυχίε, τα δικαιώματα των γυναικών, τα εργασιακά δικαιώματα, την ισότητα και άλλα πολλά. Η κυβέρνησή μας έχει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει ενεργειακά ουδέτερη μέχρι το 2030. Είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα παγκοσμίως θα έλεγα. Ούτε και για μα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Εργαζόμαστε σκληρά για να φτάσουμε εκεί. Όμως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό δεν θα υλοποιηθεί παρά μόνο μετά από συνεργασία με όλους τους τομείς, με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία των πολιτών, το δημόσιο. Πιστεύουμε πως είναι εφικτό λοιπόν, παρότι δύσκολο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, τα κεφάλαια σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, κάνατε αρκετές ερωτήσεις και από αυτές ε, κατέστησα σαφές ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική και θα συνεχίσει να είναι. Καλώς, θεωρούμε. Γι' αυτό και στην παρουσίασή μου τόνισα τον πολύ σημαντικό ρόλο της εφαρμογής της νομοθεσίας. σε ό,τι αφορά την Αφρική, την Ινδία και τις υπόλοιπες υπήρους. Οι προκλήσεις παγκοσμίως για το διεθνές εμπόριο αποδεικνύουν ταυτόχρονα την διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ όλων των θεμάτων μεταξύ της εμπορικής πολιτικής, της ε, αναπτυξιακής πολιτικής, της ανθρωπιστικής πολιτικής, των ζητημάτων ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Όλα συνδέονται. Τώρα, Ταϊβάν. Ρωτήσατε για την κατάσταση που επικρατεί και τη θέση μας. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε εξετάσει στο Συμβούλιο το ζήτημα αυτό. Και με ρωτήσατε επίσης και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα συνεχίσουμε την επεξεργασία της ιατροποποιημένης πρότασης για το θέμα αυτό τους ερχόμενους μήνες και για το ζήτημα των ε, κρατικών συμβάσεων. Επίσης, εξετάζουμε τις τεχνικές ε, πτυχές της ε, πρότασης και το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής θα φανεί τους ερχόμενους μήνες. Γι' αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα ε, να προβούμε σε εκτιμήσεις. Έπειτα, με ρωτήσατε και για τον ε, κανονισμό περί διπλής χρήσης. Καταρχάς, η νέα εκδοχή του κανονισμού θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή σε θέματα εφαρμογής και επιβολής. Θα πρέπει να δημιουργηθούν διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής και συντονισμού. Και επίσης θα πρέπει να αυξηθεί ο διάλογος με τις τρίτες χώρες έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός αυτός ο κανονισμός. Κάτι άλλο που άκουσα για την ε, προσαρμογή για την προσαρμογή στα σύνορα σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα. Πρέπει να δούμε πόσο εφικτή είναι η δημιουργία μηχανισμών τέτοιας ε, προσαρμογής, έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα ως προς τις ε, τιμές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή διότι είναι πολύ διάστατο θέμα. Γι' αυτό και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας φέτος το φθινόπωρο. Ινδία τώρα. Με την Ινδία υπάρχει ένας ε, συνεχιζόμενος διάλογος μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Όπως γνωρίζετε, η Ινδία είναι ένας ε, σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, από την άλλη, Ήδη αναφέρθηκα στην Κίνα στην παρουσίασή μου. Η Κίνα λοιπόν είναι προφανές πως είναι πάρα πολύ σημαντικός οικονομικός εταίρος. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να δούμε τι, τα ζητήματα που άπτονται των εμπορικών σχέσεών μας με την Κίνα. Αφορούν έτσι κι αλλιώς πολλούς τομείς ε, όπως εμπορική, πολιτική, εσωτερική, πολιτική, επενδύσεις κτλ. Η μεταρρύθμιση μάλιστα του ΠΟΕ θα ε, δώσει περισσότερη ασφάλεια και συμμετρία στις εμπορικές μας σχέσεις με την Κίνα. Η Κίνα θα πρέπει να κάνει τα λόγια για ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά πράξη διότι έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, γι' αυτό λοιπόν και τώρα οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε την εργαλειοθήκη μας σε ό,τι αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε και αυτές τις πτυχές. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε τις αντιπαλότητες που έχουν προκύψει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και να προσπαθήσουμε να τοποθετηθούμε σε αυτή τη σχέση των ε, τριών δυνάμεων. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχουν ζητήσει άλλοι 11 συνάδελφοι το λόγο. Ε, μπορείτε ίσως να απαντήσετε σε ερωτήσεις αυτές κατά τον δεύτερο κύκλο ερωταπαντήσεων. Τώρα, ο κάθε ένα σας έχει ένα λεπτό και ο Πίερικ έχει το λόγο. Κύριε Σχρέιπερ, και ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι από τις κάτω χώρες και στις κάτω χώρες γίνεται η συζήτηση για το Mercosur και τι σημαίνει αυτό για τις οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις. Συζητούμε για την κλιματική συμφωνία, αλλά αυτό αφορά και την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη που θα πρέπει να διατηρηθεί. Κάτι μου λείπει από εκεί. Θα πρέπει να έχουμε μία αξιολόγηση για τις συνέπειες. Γελάτε λίγο τώρα, αλλά πραγματικά αυτή η συζήτηση εξαρτάται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θα συμφωνήσουμε για το Μερκοσούρι ή όχι. Και στη δική σας Προεδρία είναι τεράστια σημασία αυτό ε, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στην παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Παρακαλώ να το κοιτάξετε αυτό, γιατί αν πάρει λάθος δρόμο, τότε θα χάσουμε το τρένο, γιατί στη συνέχεια έπονται Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και λοιπή. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το κλίμα, αλλά θα πρέπει να παραμείνει η παραγωγή τροφίμων στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να μην μα κατακλείσουν οι πολυεθνικές. Περί αυτού πρόκειται ακριβώ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπουργέ. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε ε, κανόνες με κοινέ αξίες. Και όπως υπόθηκε, το εμπόριο δεν είναι ε, η συνήθις ε, business, αλλά έχει να κάνει με τις αρχές και τις αξίες μας. Έχω ένα καλό παράδειγμα και μια πρόκληση που θα περίμενα να μας απαντήσετε. Η Τουρκία είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα για τη δυνατότητα επιβολής μας και ε, εφαρμογής. Αποτύχαμε ικτρά ως προς την προώθηση εκεί των αξιών και των αρχών μας. Πολύ σύντομα. Εξακολουθεί να κατέχει το βόρειο τμήμα της Κυπριακής ε, Δημοκρατίας η Τουρκία, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει παρά τη δέσμευσή της. Και τρίτον, πρόσφατα ε, κυριολεκτικά ε, εισέβαλε στην ΑΟΣ ε, της ε, Κύπρου με πολεμικά σκάφη και παραβιάζει έτσι τον Ευρωπαϊκό Νόμο και το Διεθνές Δίκαιο. Τι θα προωθήσει κατά της Τουρκίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ξέροντας ότι πρόσφατα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, εξήγηλε μέτρα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι κυρία Μπρικμά, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ επίκαιρα αυτά που μας λέτε, είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας ως προς το σεβασμό των κεφαλαίων της βιώσιμης ανάπτυξης βιβωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών και τώρα έχει έρθει η ώρα να επηρεάσουμε και να ε, μεταξελίξουμε αυτά τα έγγραφα έτσι ώστε τα κεφάλαια αυτά να γίνουν νομικά δεσμευτικά. Το είπατε, το υπογραμμίσατε, το τονίσατε, το στείλατε σε επιστολή στην κυρία Μογκερίνη, ακόμα και αν πρόκειται για το Μερκοσούρ. Πέρα από αυτές τις καλές προθέσεις που εμείς καλώς ορίζουμε και θα παρακολουθήσουμε πώς θα φροντίσετε ε, να γίνουν αυτά τα κεφάλαια νομικά δεσμευτικά, υποχρεωτική εφαρμογή στο μέλλον συμφωνείτε να διοριστεί ένας ε, trade officer, ένας ε, ε, αρμόδιος που θα είναι επιφορτισμένος με την επιβολή. Συμφωνείτε να υπάρχει αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επιφορτιστεί με την επιβολή αυτών ε, με ένα χαρτοφυλάκιο για το κλίμα, το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα. Επίσης, οι συζητήσεις αρχίζουν τώρα να γίνονται και στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ποιο είναι το πρόγραμμα, το σχέδιο δράσης που θα προτείνετε έτσι ώστε να επιβάλλετε την εφαρμογή αυτών. Η κυρία Κίτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου το πρωί. Αναφερθήκατε στη διάσκεψη ε, το Δεκέμβριο για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα πολύ ευπρόσδεκτη. Θέλω να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πρώτον, ε, καλωσορίζω την κοινωνία των πολιτών στη Φιλανδία, τα συνδικάτα και τις οργανώσεις των εργοδοτών. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τη βιομηχανία του καουτσούκ ε, ε, στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Ρωτώ, τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη. Πολύ συγκεκριμένο μπορείτε να κάνετε εσείς. Υπάρχουν διεθνείς διαπραγματεύσεις αυτό τον καιρό που τρέχουν στη Γενέβη για ένα δεσμευτικό σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμεί ω Ευρώπη έχουμε τα χέρια μα δεμένα γιατί δεν έχουμε διαπραγματευτική εντολή από το Συμβούλιο. Εσεί θα φροντίσετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να διαπραγματεύεται σωστά διεθνώ για να έχουμε νομικά δεσμευτική δράση, όχι απλώ λόγια για την βιωσιμότητα, αλλά συγκεκριμένη δράση και πράξη. Η κυρία Ραφαέλα, παρακαλώ. Yes, thank you. Ναι, ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αφορά την Αφρική και ελπίζω να μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα από όσα είπατε στον πρώτο γύρο. Είπατε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κείμενες συμφωνίες θα εφαρμοστούν στην Αφρική, αλλά γνωρίζουμε αρκετά για την αποτελεσματικότητα αυτών των συμφωνιών. Και επίσης ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτές τις συμφωνίες ε, η Συμφωνία του Κοτονού ε, ε, προσέφερε αυτή τη ε, δυνατότητα και πρέπει να δούμε αν μπορούμε να τους προσφέρουμε και αυτή τη δυνατότητα. Ο κύριος Γκούνας, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για το φιλόδεξο πρόγραμμα της χώρας σας αυτές τις χώρες. Ένα ερώτημα. Πρόσφατα συναντήθηκα με τον τομέα του ελαιολάδου στην Ανδαλουσία ε, στην Ανδαλουσία, η Ισπανία και η Ευρώπη είναι παγκόσμιος ηγέτης ε, στα θέματα αυτά και εξάφρι, εκφράστηκαν ε, αμφιβολίες όσον αφορά τη συμφωνία για το γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα στη συμφωνία του Μερκοσούρ. Ο τομέας αυτός εντός εισαγωγικών φυσιάζεται για να ανοίξουμε πόρτες σε βιομηχανικούς τομείς. Το Μερκοσούρ που είναι μεγάλη μας πρόκληση λοιπόν αμφισβητείται όσον αφορά τη διαχείριση της κυβέρνησης Μπολσονάρο για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και φυσικά υπήρξαν και επικρίσεις ε, για πιθανό βέτο στην επιογραφή του, αλλά και εντός της Ευρώπης υπήρχε συζήτηση για το κατά πόσον ε, και πάλι ο τομέας της Γεωργίας ε, θα υποστεί ζημίες αν εφαρμοστεί πλήρως αυτή η συμφωνία. Η Φιλανδική Προεδρία θα εγγυηθεί ε, ότι θα γίνουν σεβαστές ε, οι δυνατότητες αυτές ε, και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η κυρία Πέτρα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ως ε, υπουργό ε, Εμπορίου και Αναπτυξιακές Βοήθειες ε, μπορείτε να δείτε τι ακριβώς χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να ενταχθούν στις αγορές του παγκοσμίου εμπορίου, αλλά να έχουμε και μια αξιοπρεπή κοινωνία με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμό του κράτους δικαίου και φυσικά σεβασμό και περιβαλλοντικών προτύπων. Η ερώτησή μου αφορά την συμφωνία ε, ε, για τις επενδύσεις. Ε, ξέρουμε ότι είναι καλογραμμένη, αλλά ξέρουμε ότι η Νότια Κορία μετά από 8 χρόνια δεν έχει υπογράψει. Και ξέρω ότι μια χώρα μπορεί να μην αποτελεί και υπόδειγμα για τις υπόλοιπες, αλλά ε, μήπως στη διάρκεια της Προεδρίας σας θα δούμε τα κεφάλαια αυτά και είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και μπορούμε να δούμε και ποιος θα διαπραγματευτεί όταν υπάρξουν προβλήματα. Και θα ολοκληρώσω στα φιλανδικά. το εξάμεινο της ε, Φιλανδικής Προεδρίας. Ελπίζω να πάει καλά και να θριαμβεύσουμε και ελπίζω στη διάρκεια του εξαμήνου μας ε, να μην ε, διακοπεί καμία διαπραγμάτευση ε, και να συνεχίσουν να είναι ανοιχτέ ε, οι πόρτε διαπραγμάτευση και με το Μερκοσούρ και με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε να διακοπούν οι διαπραγματεύσει αυτέ στη διάρκεια του εξαμήνου μα και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στα στάδια αυτά. Η κυρία Σιμακοπούλου, Πρόεδρε, Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ούσουλα Φοντερ Λάιεν μας μίλησε για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρή Ευρώπης στον κόσμο και ιδιαίτερα για την ενίσχυση της Ευρώπης ως παγκόσμιο ηγέτη και εκείνο που θέτει τα πρότυπα, τα στάνταρ για ένα ισχυρό ανοιχτό εμπόριο. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις, μια διπλή ερώτηση. Πώς συνδέονται με τις προτεραιότητες κυρίας Φοντερ οι φιλανδικές προτεραιότητες. Και δεύτερον, ποια είναι η στρατηγική μας προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, που ε, συμφωνεί η κυρία Φόντερ Λάιεν να αρχίσουν διαπραγματεύσει με τις κυβερνήσεις των Σκοπίων και των Τυράννων. Έχετε καμία ειδική έτσι, χρονική ε, προσέγγιση, κυρία Κατάινε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε Υπουργέ Σκινάρη, είναι μεγάλη περηφάνεια για μένα ο Υπουργό Φιλανδία να λέτε ότι το εμπόριο πρέπει να βασίζεται στι αξίε, στου σωστού κανόνε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Φιλανδική Προεδρία επισημαίνει για άλλη μια φορά τη σημασία των κανόνων του παιχνιδιού. Ε, κάτι ε, το οποίο δεν αρκεί να το επαλαμβάνουμε συνεχώς. Όσε φορέ και να το επαναλάβουμε, δεν φτάνει. Ε, με τι Ηνωμένε Πολιτείε ε, το, ε, την Άνοιξη ήταν μεγάλο το σοκ όταν διακόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις με Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα και είναι τόσε μεγάλες οι εντάσεις, ιδιαίτερα σε καιρούς σαν αυτούς και πλησιάζουν και τα όσα επιβάλλει ο κύριος ε, Τραμπ ε, ε, και είναι και πρώτον πυλών τα θέματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. κυρία Μουνιώθ, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, η κυρία Πινιέρο ε, για την καθυστέρηση. Παρακολουθούσα όμως τη συζήτηση μέσω web streaming. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να αναλάβουμε τα ενία ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική επιρροή. Γι' αυτό ακριβώς και οι εμπορικές διμερείς σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν δεν μπορέσουμε όμως να εγγυηθούμε κατάλληλη εφαρμογή των αρχών και αξιών που υπερασπιζόμαστε μέσω αυτών των διμερών συμφωνιών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτήσουμε την επιρροή που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς και θα ήθελα να ξέρω πώς μπορείτε να δώσετε όθηση για μεγαλύτερη ε, εφαρμογή των συμφωνιών. Υποστηρίζω απόλυτα την πρόταση της συναδέλφου Κίρτον Ντάρλινγκ όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου και τη σημασία της κατάλληλης εντολής ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση μιας δεσμευτικής ε, συμφωνίες για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσον αφορά τις σχέσεις με την Λατινική Αμερική θα ήθελα να ξέρω αν θα προωθήσετε την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Μεξικό και τη Χιλή και για την διπουργική ε, διάσκεψη του ΠΟΕ τον ερχόμενο Ιούνιο τι στόχους ε, έχετε. Ευχαριστώ. Η κυρία... Thank you, Minister. I'd hope to be... Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το Μερκοσούρ και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά δεν θα ήθελα να φύγετε με κάποια παρανόηση από την αίθουσα αυτή για την κατάσταση στη Βρετανία. Συμφωνείτε λοιπόν με το μεγαλύτερο τμήμα του Βρετανικού πληθυσμού ότι το χειρότερο σενάριο για το Brexit, ε, ε, πολύ χειρότερο από την ε, σκληρή συμφωνία, θα ήταν μια συμφωνία χωρίς, μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία και αυτό είναι ε, ανεύθυνο και επικίνδυνο και έχετε κάτι για μια στρατηγική διαπραγμάτευση, για μια τέτοια ή οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση εμπορίου που βασίζεται σε μπλόφες ε, και επιδείνωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, πάψει να είναι ένα σοβαρό και αξιοσέβαστο εμπορικό εταίρο, όχι μόνο με, το με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλου ε, παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Υπήρξαν πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και είμαι βέβαιος ότι το προσωπικό σας ε, σημείωσε όλες τις ερωτήσεις και ίσως θα μπορούσε να στείλει ίσως και κάποιες ε, γραπτές απαντήσεις, αλλά ε, να σας δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση από τον συνάδελφο της κατοχώρες. Προσπάθησα να ακούσω στα Ολλανδικά, γι' αυτό χαμογέλασα. Ε, Δυστυχώ τα Ολλανδικά μου είναι κάπως κουριασμένα. Με συγχωρείτε. Ε, να σας απαντήσω όμως ε, σε ό,τι αφορά την Γεωργία και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Τα αποτελέσματα για το κομμάτι της συμφωνίας που αφορά τη Γεωργία είναι λογικά, είναι ισορροπημένα. Η συμφωνία μάλιστα θα δώσει νέες ευκαιρίες για εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα θα προστατεύσει ορισμένους ευάλωτους τομείς με ε, δασμολογικές ποσοστώσεις, με χρηματοδοτική στήριξη μεταξύ άλλων. Επίσης θα προστατεύονται και ορισμένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία λοιπόν δεν θα αλλάξει τους ε, κανόνες περί ασφάλειας των ε, τροφίμων, μάλιστα θα τους ενισχύσει. Και θα ενισχύσει επίσης τη διαφάνεια σε πολλούς τομείς. Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζουμε τις ε, ανησυχίες πολλών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αλλά η συμφωνία περιέχει πολύ ισχυρές διατάξεις για τις οποίες θα δεσμευτούν και οι δύο πλευρές, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσω της Συμφωνίας να συνεργαστούμε με τις ε, χώρες Mercosur για περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι η απαγόρευση εισαγωγή βόλιου κρέατο και άλλων προϊόντων από τη Βραζιλία είναι κάτι το εφικτό προ το παρόν. Φυσικά η κατάσταση στην περιοχή του Αμαζονίου επιδεινώνεται και θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση όλων των ε, δυνατοτήτων που έχουμε για να επιληθεί αυτή η κρίση. Επίσης, η απελευθέρωση του γεωργικού εμπορίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ε, συμφωνία σε ένα ευρύτερο όμω πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι σταδιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόηο κρέας από 99.000 τόνους αποτελεί λιγότερο από το 1% της συνολικής παραγωγής βόηου κρέατος της Βραζιλίας, το οποίο η οποία ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, ανταγωνιστικότητα, είναι πολύ σημαντικό σημαντικό στοιχείο για την ε, Προεδρία μας και φυσικά η Προεδρία της ε, Φιλανδίας τονίζει την ε, σημασία που πρέπει να έχει η έρευνα και η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ηγετική θέση της Ευρώπης στον χώρο αυτόν. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την Τουρκία. Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση και υπάρχουν ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα αυτό αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η ερώτηση σχετικά με την ε, Γεωργία. Να επαναλάβω ότι η Γεωργία δεν συμπεριλαμβάνεται στην ε, διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να απαντήσω στην ερώτηση για την ομιλία της Ursula von der Να πω ότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, μισό λεπτό να τις κοιτάξω ξανά. Να πω λοιπόν ότι η Ursula von der τόνισε τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών, όπως και η κυβέρνησή μας το έκανε. Συμμεριζόμαστε λοιπόν ε, τις επεπιθήσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν στο έπακρο. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις. Θα μπορούσα βέβαια να συνεχίσω και να απαντήσω σε όλες, αν θέλετε. Είμαι σίγουρος. The binding treaty. Yes. And actually Africa. Ναι, ναι, η δεσμευτική συνθήκη. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε ο κύριος Υπουργός. Ναι, Αφρική, το ξέχασα. Η κυβέρνησή μας λοιπόν έχει δεσμευθεί ε, για την κατάρτιση μιας στρατηγικής για την Αφρική, διότι θεωρούμε πως η Αφρικανική Πύρος είναι πολύ σημαντική ε, και θα είναι μελλοντικά όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ανέφερα, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο εμπόριο, στην αναπτυξιακή βοήθεια και το εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στην ε, Αφρική, στον χώρο των πορείου και της ε, ανάπτυξης. Θα υπάρχει λοιπόν μια κοινή προσέγγιση. Αυτά νομίζω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Βλέπετε, φαντάζομαι, ότι η Επιτροπή μας είναι πολύ δραστήρια και όλοι μας έχουμε επίγνωση της μεγάλης πρόκλησης που βρίσκεται ενώπιόν μας και θέλουμε να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου με την ε, Φιλανδική Προεδρία έτσι ώστε στο τέλος του χρόνου να ε, έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρώπης αλλά και για τις χώρες εταίρους μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και καλή τύχη στην Προεδρία σας. Okay. You will continue. One yeah. more picture. One more picture. So. He's my special advisor, young but very talented okay, good. okay. Thanks. So, dear colleagues, now... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την πρώτη μας ψηφοφορία στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. And according to the rules, uh... Και σύμφωνα με τον κανονισμό μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τώρα την ηλεκτρονική δυνατότητα. Αλλά όχι, η γραμματεία μου λέει δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες επισημότητες, διότι δεν είναι τελική ψηφοφορία. Μόνο τέσσερις ε, τροπολογίες έχουμε να ψηφίσουμε. Άρα τούτη τη φορά δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, προτείνει η κυρία Χιούμπνερ να κάνουμε ένα τσεκ, έναν έλεγχο, όχι μόνο εάν μπορείτε εσείς να ψηφίσετε, αλλά εμείς θα τσεκάρουμε και τη δύναμη των πολιτικών ομάδων και αν εκπροσωπήσετε σωστά. Λοιπόν, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. And, uh, the vote is open. Και αρχίζει τώρα. Members here and the vote is open. 41 μέλη είναι παρόντα. <laughs> Τι είναι, καλοκαίρι ή χειμώνα, τι ψηφίζουμε. Δεν δουλεύουν τα μηχανήματα ή για ποιο λόγο ζητήσατε το λόγο. Α, έχουμε πρόβλημα. 41 μέλη έχουμε παρόντα με κάρτες και ε, δεν δουλεύει. Α, είναι λάθος όνομα λέει ε, α, έτσι κι αλλιώς περισσεύει ένας από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ωραία, βγάζω εγώ τη δική μου κάρτα τότε, λέει ο πρόεδρος. Okay, now we have 39 members. 39 τώρα. Και η Χάιντι που δεν έχει κάρτα, Χάουταλα. Και εσείς έχετε λάθος όνομα εκεί, αλλά Τώρα δεν έχει σημασία το όνομα, έχει σημασία το νούμερο. Δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, όλα εντάξει, έχουμε αρκετά μέλη για να ψηφίσουμε. Όχι ηλεκτρονικά, τάσω σχήρως. Έχουμε την πρώτη τροπολογία για τη γραμμή 3042 του προπολογισμού ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η δεύτερη τροπολογία γραμμή 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τρίτη τροπολογία 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τέλος έχουμε μια τροπολογία στο κονδύλι 16030104, μια συμβιβαστική τροπολογία που έρχεται να αντικαταστήσει την αρχική. Ψήφι υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Αυτή ήταν η σύντομη ψηφοφορία μας, πρώτη στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία και έληξε. Ευχαριστώ. Αν θέλει να φύγει κάποιος τώρα από αυτή την καταπληκτική συνεδρίαση και την καταπληκτική μας επιτροπή, να το πράξει παρακαλώ ησύχω. Then we switch to point 10, dear colleagues. It's a presentation of... Σημείο 10. Παρουσίαση ε, της έκθεσης για τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Έκθεση για το έτος 2018. Ξέρετε ότι είναι ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ επικοδομητική έκθεση πιστεύω πάντα που περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίω στο εμπόριο. Για οι ε, φραγμοί εμπορικοί κοστίζουν πάρα πολύ φυσικά και σε αυτόν τον κόσμο που είναι σήμερα γεμάτος προκλήσεις είναι πολύ οι και τα εμπόδια, ιδιαίτερα στην Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αλλά εκτός αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εξαλείψει 35 τέτοιους εμπορικούς φραγμούς το 2018. Και αυτό θα είναι τμήμα της έκθεσης που θα μας παρουσιαστεί. Θέλω να δώσω το λόγο στον Φρανσίσκο Πέρι Κανάντο που εκτελεί χρέη διευθυντού στην αρμόδια διεύθυνση. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Αγαπητοί κύριοι, αγαπητές κυρίες, με μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω τις σημαντικότερες πτυχές της έκθεσης για τους εμπορικούς και επενδυτικούς φραγμούς την ολοκληρώσαμε μέσα στο καλοκαίρι και όπως γνωρίζετε η αγορά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, πυλώνας. Η επόμενη επιτροπή θα έχει το θέμα αυτό ως ύψιστη προτεραιότητα, διότι δίχως αυτό δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε παρουσίαση πρέπει να ε, ξεκινήσει και να τελειώσει με τον ίδιο ε, τρόπο και αυτό ακριβώς ε, θα κάνω. Αρχικά, να σας ε, πω ότι ο προστατευτισμός αυξάνεται και ε, δεν βλέπουμε να αλλάζει αυτό στο μέλλον. Έπειτα, η στρατηγική μας για την αγορά θα δώσει αποτελέσματα, θα ε, αρθούν οι φραγοί, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές. Για τις αλλαγέ λοιπόν χρειάζεται δουλειά. Για να έρθουν οι φραγμοί χρειάζεται δουλειά. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μας, ε, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό. Θα σταθώ λοιπόν στην παρουσίασή μου σε αυτούς τους τρεις ε, τομείς. Στην Επιτροπή υπάρχουν αρκετά νέα μέλη. Θα σας εξηγήσω λοιπόν αρχικά για ε, την ε, στρατηγική ε, πρόσβαση στην αγορά. Είναι μια στρατηγική που αρχίζει από τη βάση προς τα πάνω και στόχο έχει να έρθουν οι φραγμοί σε όλους τους τομείς εμπορικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των επιχειρήσεων, των σχετικών οργανώσεων και των κρατών μελών για να δοθεί μια στρατηγική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μέτρα Φυσικά, αυτό θα ωφελήσει περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πιο ευάλωτες δηλαδή. Και η εμπειρία μας από το περασμένο έτος επιβεβαιώνει αυτήν την ε, άσχημη τάση της αύξησης των φραγμών στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Και μάλιστα αν κάνουμε μία σύγκριση ε, ανά τα έτη θα δούμε ότι πέρυσι οι φραγμοί αυτοί αυξήθηκαν κατά πολύ. Υπάρχει περισσότερη εμποροκρατία, περισσότερος προστατευτισμός και αυτό μας ε, δείχνει ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε και να ξεκινήσουμε δουλειά έτσι ώστε να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τους φραγμούς αυτούς με όποιον τρόπο μπορούμε. Οι φραγμοί αυτοί επηρεάζουν πολύ σημαντικά τις εξαγωγές μας, μας κοστίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και ε, εστιάζουν σε, στον αντίκτυπο και στους εμπορικούς εταίρους. Σκεφτείτε τις Ηνωμένε Πολιτείες, δεν σας εκπλήσει αυτό νομίζω. Σκεφτείτε τι έχει γίνει με τον χάλιβα και το αλουμίνιο. Ε, από την άλλη, Κίνα, ε, τα μέτρα στον κυβερνοχώρο που επηρεάζουν τις ε, τεχνολογίες επικοινωνίας και ε, πληροφορίας. Και Ινδία με τα γεωργικά προϊόντα, το δέρμα, ε, τα καλλιντικά. Τώρα, η Αλγερία είναι ένας επέκτης που ίσως σας ξαφνιάσει. Όμως η Αλγερία έχει λάβει ένα σύνολο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει μέχρι και απαγόρευση εισαγωγών ορισμένων προϊόντων. Αυτό έχει πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Μάλιστα, η περιφέρεια της ε, Μεσογείου έχει επηρεαστεί κατά πολύ περισσότερο από ό,τι έχει επηρεάσει η Κίνα την, ε, το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, περιοχή αυτή μάλλον. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται από ε, την ε, μεταλλουργία, την ε, πληροφορική και την τεχνολογία. Νομίζω πως οι επιπτώσεις είναι αισθητέ. Πρώτον από την στρατηγική της Κίνας, μετά από τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ινδίας και της Αλγερίας. Και τις επιπτώσεις αυτές θα τις νιώθουμε για πολύ καιρό ακόμα. Καταρχάς, ε, να πω ότι αυτά που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά έχουν ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια. Ε, πριν από δύο χρόνια, λοιπόν, πιάσαμε δουλειά και εστιάσαμε σε τρεις τομείς. Πρώτον, στο συντονισμό με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη-μέλη για συντονισμένη δράση. Μέσω των πρεσβειών μας στις τρίτες χώρες θα καταφέρουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έπειτα, επιλέξαμε να δώσουμε προτεραιότητες, να τις ιεραρχήσουμε. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα ταυτόχρονα, γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να εστιάσουμε στις προτεραιότητες και στις πιο εφικτές λύσεις. Έπειτα, ευαισθητοποίηση μέσω διαφόρων εκδηλώσεων για την ε, αγορά. Έχουμε εστιάσει σε έξι κράτη-μέλη, στα οποία έχουν γίνει τέτοιες εκδηλώσεις. Τους επόμενους 18 μήνες θα γίνουν εκδηλώσεις σε άλλα έξι, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, να γνωρίζουν ότι υπάρχει μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εκεί για να τους βοηθήσει, για να έρθουν οι φραγμοί. Και νομίζω πως αυτή η προσέγγιση μας έχει βοηθήσει στο να εντοπίσουμε τους μεγαλύτερους ε, κινδύνους, τους μεγαλύτερους φραγμούς. Έπειτα, όπως ε, είπαμε και νωρίτερα, έχουμε ε, βοηθήσει να εξαλειφθούν 35 τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί το τελευταίο έτος σε πολλούς τομείς Αλλά οι τομεί που επωφελήθηκαν περισσότερο είναι από τη μία η αυτοκινητοβιομηχανία, μετά ο γεωργικό τομέα ε, και ο τομέα των τροφίμων και ε, ο τομέα των καλλιτικών προϊόντων. Αυτοί είναι οι τομεί που επωφελήθηκαν περισσότερο από την ε, περσινή μα δραστηριότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι χώρε τι οποίε εστιάσαμε, καλύπτουμε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος και ε, θα σταθούμε τώρα στην Αίγυπτο, στην Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, την Νότια Κορέα. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν έχουμε άρει πολλούς σημαντικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, αν θυμάστε, μας ε, δώσατε αρκετή δουλειά για το σπίτι και ένα από αυτά που έπρεπε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε ποιο είναι το όφελος της άρσης των φραγμών στις εξαγωγές μας. Έγινε λοιπόν μία εκτίμηση της κατάστασης και τώρα σε αιτήσια βάση διενεργούμε ε, τέτοιες εκτιμήσεις. Γι' αυτό λοιπόν από το 2014 μέχρι το 2017 η άρση των φραγμών μας οδήγησε σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κέρδος. Δεν είναι άσχημα αυτά. Έπειτα, το δεύτερο που μας είπατε να κάνουμε είναι να δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν την απασχόληση. Αυτό ήταν πιο δύσκολο. Δεν καταφέραμε να το αναλύσουμε λεπτομερώς, όμως με βάση τους υπολογισμούς μας, οι εξαγωγές απασχολούν 36 εκατομμύρια εργαζόμενους. Έχουμε λοιπόν άλλα 6 ε, περίπου δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον τα οποία αναλογούν σε 100.000 ε, θέσεις εργασίας επιπλέον. Και μιλάμε για θέσεις εργασίας οι οποίες ε, βρίσκονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια κάποια ικανοποίηση ως αποτέλεσμα που επιτύχαμε, όμως ας ε, μην είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Η Κίνα είναι ένας πολύ δύσκολος ε, εταίρος, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το κάνουμε αυτό από πέρυσι. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας απέναντι σε αυτό το τόσο μερκαντιλιστικό κράτος και να εστιάσουμε στην ε, προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια στο εμπόριο σε όλους τους ε, τομείς της πολιτικής. Πρέπει να επιμείνουμε στην ε, πρόσβαση στην αγορά. Και θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που έχουμε είναι η θέση του υπεύθυνου επιβολής. Κάτι που η κυρία Φοντερ Λάιεν αποκάλυψε ήδη στη, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της. Χρειάζεται βεβαίω και ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση. Νομίζω πω εδώ έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότερε μικρομεσαίες επιχειρήσει για το τι κάνουμε. Τέλο, ο θεμελιώδη ουσιαστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσεί μπορείτε να ε, μα ε, βοηθήσετε σε αυτό το δύσκολο έργο με πολλού τρόπου. Όσοι ήσασταν εδώ και στην προηγούμενη θητεία θα θυμάστε ίσως ότι οι ευρωβουλευτές είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της εμπορικής πολιτικής που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Είστε φορείς μεγάλης αξιοπιστίας, ιδιαίτερα απέναντι σε τρίτες χώρες. Να σας ε, θυμίσω ότι τον αντίκτυπο που είχατε στην επίσκεψη στο Πεκίνο. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι αντιπροσωπείες που έχετε, που στέλνετε σε τρίτες χώρες και η πίεση που ασκείτε πολιτικά για την άρση των ε, φραγμών αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε στα χέρια σας μεγάλη επιρροή και πρέπει να την ασκήσετε. Αυτό από τη μία είναι ε, ένα κομμάτι της συνεισφοράς σας. Από την άλλη, νομίζω πως μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά ενημερώνοντας. Ο αξιότιμος κύριος Λαντσίνη έχει αποχωρήσει από την αίθουσα και ήθελα να τον επενέσω διότι πριν από μερικούς μήνες διοργάνωσε μια εκπληκτική εκδήλωση στη Λομβαρδία για την πρόσβαση στην αγορά. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η διοργάνωση εκδηλώσεων νομίζω πως μπορεί να έχει μεγάλα αποτελέσματα Αυτά λοιπόν ε, προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ο δρόμος θα γίνει ακόμα δυσκολότερος, όμως θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι μας, οι πολίτες θα πρέπει να είναι σίγουροι για αυτό που κάνουμε εμείς, ότι έχουμε ένα σχέδιο για να γίνει πιο αποτελεσματική καταπολέμηση των φραγμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως φαίνεται να υπάρχει φως ε, στην άκρη του τούνελ. Αυτό είναι καλό. Και τώρα να περάσουμε στα μέλη. 1,5 με 2 λεπτά θα έλεγα. Και η κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο. Ε, είμαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα έκανε και την παρουσίαση της έκθεσης. Ήθελα να θέσω δύο πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Είπατε και όντως ισχύει αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό δυστυχώς ε, ε, τι γίνεται με την πολιτική της ε, Αλγερίας για δασμούς και άλλους μη δασμολογικούς φραγμούς. Στην περιοχή της Βαλένθια είναι, έχουμε την πρώτη χώρα παραγωγό ε, κεραμικής και εξαγωγές κεραμικής και τι γίνεται με την ε, με τα ναι, εξαγωγή κεραμικών. Άλλαξαν πολύ τα πράγματα λόγω της αλλαγής της τάσης Αλγερίας. Υπάρχει συμφωνία, είναι πολύ λεπτή η κατάσταση και θα ήθελα να ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτού. Δεύτερον, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ε, έχουμε ένα ακόμα στοιχείο ε, εμπορικών φραγμών και γι' αυτό οι νέες συμφωνίες της νέας γενιάς συμπεριλαμβάνονται και τα θέματα των δημοσίων συμβάσεων. Εγώ όμως στις αναφορές που έκανα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες ε, για τις περιοριστικές ε, διατάξεις και τα όσα γίνονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να υποδοθούν και να έχουμε κάτι καλύτερο. Πώς θα βελτιωθούν τα πράγματα λοιπόν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα έκθεση και την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το κείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην Ινδία. Μόλις έβαλε ένα νέο φορολογικό ε, σύστημα για τη φορολόγηση ε, επενδύσεων ε, χαρτοφυλακίου από το εξωτερικό. Τι γίνεται διεθνώ με τη φορολογική πολιτική και εδώ αναφέρομαι και στι ΗΠΑ και σε άλλους εταίρους. Επηρεάζει αυτή άμεσα την πρόσβαση στην αγορά. και για τα αγαθά και για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις μάλλον τις ξένες στις τρίτες χώρες. Αυτό είναι φραγμός ή όχι. Όταν μιλάμε για το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν και τις δικές τους εγχώριες οικονομίες οι διάφορες χώρες. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το πώς οργανώνουμε την ε, ε, αλυσίδα παραγωγής αξίας. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη ερώτηση και ε, στη χάρτα την ενεργειακή. Κατά κάποιο τρόπο και αυτό Ε, επιτίθεται στα κρατημέλη και δεν τα αφήνει να αναπτύξουν την εναλλακτική τους ενεργειακή πολιτική. Όταν συζητούμε για την κατάσταση ε, της παλιάς παραγωγής ενέργειας με νέα, ανανεώσιμες κτλ. Με την ηλιακή και άλλες ανανεώσιμες. είναι και αυτό ένα εργαλείο που δρά περιοριστικά ως φραγμός ε, στην ανάπτυξη νέων ε, βιομηχανικών και ενεργειακών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, στη δωρηνή συζήτηση για τις επενδύσεις στην πολυμερή έχουμε ένα πρόβλημα. Και τον Απρίλιο, το είδαμε, ήρθε μια πρόταση που θεωρήθηκε ευκαιρία αλλά πολλές φορές οι επενδυτές ε, ε, έχουν ε, αυξημένα δικαιώματα απέναντι στα κράτη και στις λήψεις αποφάσεων και στις δικαστικές αποφάσεις. Πώς θα λυθεί αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Warborn. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ευχαριστώ για την πολύ καλή έκθεση. Έχω δύο ερωτήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Για την Κίνα και τους νέους φραγμούς, στην έκθεση λέγεται και παραθέτω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις απαιτούν περισσότερο ε, προσπάθειες πολύ καλά συντονισμένες για να βελτιώσουμε την πρόσβαση της αγοράς ε, σε θέματα ε, εμπορίου με την Κίνα. Ποια είναι καλά παραδείγματα προσπαθειών για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, επειδή η έκθεση βασίζεται σε έρευνα ε, στο χαμηλότερο επίπεδο. Μας ε, λέτε ότι πρέπει να ενημερωθούμε περισσότερο. Έχετε κάποια εικόνα ε, ε, για τους φραγμούς που δεν γνωρίζουμε και δεν αναφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Σαιαπύρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι νέο μέλος εδώ στην Επιτροπή ε, και έχω ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσατε για συνειδητοποίηση από πλευράς κοινοβουλίου. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά έχετε καμιά πρόταση πιο συγκεκριμένη. Γιατί απλώς μια παρατήρηση είναι. Και πρέπει να πω ότι το θέμα του Μερκοσούρ φέτος το καλοκαίρι μου έκανε τεράστια εντύπωση σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις ε, κάτω χώρες. Είναι διοξίδιο του άνθρακα, ε, αυτό που συζητάνε είναι οι δασικές πυρκαγιές. Δεν προβάλλονται αρκετά τα θετικά από τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Εμείς δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα προδραστικά, δηλαδή εκ των προτέρων και όχι να αρχόμαστε να αντιδρούμε. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά στρέφομαι και προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από δύο-τρία χρόνια ε, είχαμε τότε τον Επίτροπο Γεωργίας ακόμα, τον κύριο Χόγκαν, ε, που έκανε μια μεγάλη εμπορική συμφωνία με την Κίνα και τον Καναδά. Και εκεί δεν εδέησε να απαραστεί ο Ολλανδός Υπουργός Γεωργίας. Δεν ενδιαφερόταν για αυτά τα θέματα. Μα αν υπάρχει μια χώρα που έχει τέτοιο εμπόριο με αγροτικά προϊόντα, αυτή είναι η Ολλανδία. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να μην υπάρχει αυτή η αρνητική προσέγγιση απέναντι σε θέμα του εμπορίου. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις γενναιόδερες παρατηρήσεις, για τη σημασία των Ευρωβουλευτών ε, για τη μείωση των εμπορικών φραγμών. Αλλά αν ε, δούμε τη ε, σελίδα 2 για τις διπλωματικές ε, δράσεις, δεν υπάρχει καμία παρουσία ευρωβουλευτών σε αυτό τον σχετικά πλήρη κατάλογο σημαντικών φορέων. Ίσως θα έπρεπε να το προβάλλετε λοιπόν και αυτό, να μην φαίνεται απλώς στο, στο παρασκήνιο. Από ό,τι κατάλαβα, αναδύεται μία εμπορική διαφορά μεταξύ ε, της χώρες παραγωγών φινικελαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πού βρίσκεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Από ό,τι κατάλαβα, κάποιες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ήδη προσφεύγουν στον ΠΟΕ για την μη χρήση του φινικελαίου ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι άποψη έχετε εσείς για αυτή την υπόθεση σε σχέση με τη ε, συμφωνία που συνάφθηκε με τον πρόεδρο Γιούγκερ και τις Ηνωμένε Πολιτείες το 2018. Ας την αποκαλέσουμε Ε, μια τροχοπέδη ώστε να μην ε, ξεκινήσει εμπορικός πόλεμος και να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Από ό,τι κατάλαβα, τμήμα αυτή τη ενδιάμεση συμφωνία ήταν ε, να διευκολύνουν τις εισαγωγές σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ω αντίφαση σε σχέση με τι πολιτικέ μα με την Νοτιοανατολική Ασία για το φινικέλαιο. Πώς βλέπει λοιπόν η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τη κατάσταση αυτή. Ο Φρανσίσκο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις θα σας παραπέμψω και στις παρουσιάσεις που θα γίνουν αργότερα στη διάρκεια της ημέρας από τις συναδέλφους ε, για ε, συγκεκριμένα θέματα. Η ερώτηση για την Αλγερία καταρχάς. Η κατάσταση βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τον ε, τομέα της κεραμικής ε, και είμαστε σε επαφές σχεδόν καθημερινά για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια πολύ καλή απόδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η Αλγερία είναι μια χώρα που έχει σαφή οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και μπορεί να μην ακολουθεί κατά γράμμα τη συμφωνία, τη διμερή συμφωνία σύνδεσης που έχουν μαζί μας. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε κάθε διπλωματική οδό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, αλλά φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο να εξετάσουμε ε, και προσφυγή σε επίλυση διαφορών βάσει της συμφωνίας. Και μάλιστα ε, εδώ πρόκειται και για ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές ε, συνέπειες. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν υπέψη και να αντιμετωπιστούν. Αυτό που κάναμε την προηγούμενη χρονιά ήταν να προσπαθήσουμε να συντονιστούμε ε, στενότερο σε κάθε κράτος μέλος αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με το εμπορικό και το πολιτικό σκέλος. Διότι Κάποιε πιο εύρωστε, αν θέλετε, εμπορικέ δράσει μπορεί να μην είναι πάντα βάση και της πολιτικής σκοπιά ε, και ε, δεν ευθυγραμμίζονται με τους ευρύτερους πολιτικούς στόχου που έχουμε με κάποιου από του εταίρους μας. Ε, πέραν αυτού βεβαίω, μπορώ να σας πω ότι εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα διότι ο αντίκτυπο για πολλού από του κλάδους μα, όχι μόνο για την κεραμική αλλά για παράδειγμα το χάλιβα ο αντίκτυπος των αλγερινών ε, περιορισμών ε, είναι πολύ σημαντικός. Ε, ο συνάδελφος Μάτε μου ψηφιρίζει να μην ξεχάσω και τα αυτοκίνητα. Δεν θα τα ξεχάσω λοιπόν τα αυτοκίνητα όταν θα σας μιλήσω για το θέμα αυτό. Τώρα, δημόσιες συμβάσεις. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα με τεράστιες ευκαιρίες ε, τη τάξη των τρισεκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις μας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, διότι πολλοί από τους εταίρους με τους οποίους έχουμε προβλήματα δεν είναι μέλη τη συμφωνία ε, ε, Κυβερνητικών Προμηθειών στον ΠΟΕ και πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ οδούς και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Επιτόπου, ε, βοηθήσαμε μια σλοβενική επιχείρηση στη Βραζιλία, παρά το γεγονό ότι δεν υπήρχε κάποια υποχρέωση από ε, πλευρά Βραζιλίας, αλλά με την παρέμβασή μας βοηθήσαμε και εξετάζονται ως υποψήφιοι σε μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα προσοδοφόρα ε, σύμβαση, χάρη σε διπλωματικές ανταλλαγές. Αυτά είναι πράγματα που δεν μαθαίνετε. Αυτό είναι, αυτός είναι ο ένας διάβλος. Ο δεύτερος διάβλος έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, στο ρόλο του ως ε, συνομοθέτης, στη συναπόφαση. Χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία προκειμένου να προστα... προβάλλουμε το πόσο ανοιχτοί είμαστε σε δημόσιες συμβάσεις. Γι' αυτό και ακριβώς το εργαλείο κυβερνητικών συμβάσεων είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι από τότε που ασχολούμαι με τα θέματα της Κίνας, ε, το γεγονός και μόνο ότι ε, το συζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς το αναφέραμε, ε, δημιουργούσε πολλή συζήτηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα εμπορικά χαρτιά, κυρίες και κύριοι, και παρακαλώ ε, να προσφέρετε στους ε, ε συναδέλφους αυτά τα, εμπορικά χαρτιά, γιατί αυτά είναι ε, αυτά τα οποία προσφέρονται σε αυτές τις ευκαιρίες. Τώρα, για την ενέργεια και τις επενδύσεις θα σας παραπέμψω στους συναδέλφους που θα έρθουν εδώ αργότερα και θα συζητήσουν τα θέματα που αναφέρατε. Όσον αφορά την ε, φορολόγηση στην Ινδία και αν αυτή είναι διάκριση για τη φορολόγηση, αυτό βεβαίως ε, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό εμπορικό φραγμό, αλλά εξαρτάται από την περίπτωση. Και πράγματι, σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ σαφείς αναπτυξιακοί στόχοι, οι οποίοι ε, υφέρπουν πίσω από αυτή τη φορολόγηση, η προσπάθειά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν χωρί να παρακολύσουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αντίθεση με τους κανόνες. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για την εξαγωγή αγαθών. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ευθύνη μας να εξετάσουμε ε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργαζομένους μας πρώτον και κυριότερον, λαμβάνοντας πλήρως ε, υπόψη και τους πολύ λογικούς ε, στόχους ανάπτυξης των υπολείπων. Υπήρχε και μια ερώτηση για το τι κάνουμε για την Κίνα και πώς πάνε τα πράγματα καλύτερα. Υπάρχουν κάποια μικρά πραγματάκια, αλλά και πολύ μεγάλα πράγματα. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά όλα τα πλήκτρα του πιάνου για να μπορέσουμε να άρουμε τους φραγμούς. Δύο παραδείγματα. Έχουμε ενισχύσει το συντονισμό επιτόπου μεταξύ των πρεσβειών ώστε να μπορέσουμε να βλέπουμε επιτόπου, για καλή, ε, παράδειγμα, ποια υπουργεία πρέπει να πιέσουμε για να αποκτήσουμε ε, αποτελέσματα για την πρόσβαση στι αγορές. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δελεαστικό, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπετε, αλλά μας επιτρέπει να έχουμε κάποιε περαιτέρω πληροφορίες και να μπορούμε να έχουμε μια αναλυτική, στρατηγική, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας που είναι πολύ καλή. Αυτό είναι το μικρό. Και τώρα να μιλήσουμε για τα σημαντικά. Και τα πολιτικά στοιχεία. Στην τελευταία σύνοδο για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια συμφωνήσαμε σε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο περιλάμβανε και μια σαφή συμφωνία από κινέζικης πλευράς για να εξετάσουν το θέμα της άρσης των ε, φραγμών στην πρόσβαση των αγορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κίνα, διότι για αυτά τα θέματα χρειάζεται υποστήριξη Τη ηγεσία για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με όλα τα τερτύπια ε, και τις δυσκολίες ε, της επαφής μεταξύ των Υπουργείων και των ε, κατώτερων στρωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει και η πρακτική δουλειά αλλά και τα πιο πολιτικά πράγματα. Με θέσετε και με ερώτηση που ξέρετε ότι δεν μπορούσα να απαντήσω. Μου άρεσε, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω κάποια σχόλια. Αν γνωρίζουμε Πώ το είπε ο τα γνωστά άγνωστα, τους γνωστούς αγνώστους κλπ. Ε, δεν τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι χάρη στην ενίσχυση της ενημέρωσης υπάρχει αύξηση στον αριθμό των ερωτημάτων που λαμβάνουμε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις χώρες που επισκεφτήκαμε. Παρεμπιπτόντως η Σουηδία υποτίθεται ότι είναι επόμενη στις επισκέψεις μας. Αυτό λοιπόν προς εσάς. Τώρα, το Μερκοσούρ. Ε, ποτέ δεν ε, μου άρεσε περισσότερο ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ερώτησή σας. Ξεχνάμε ότι σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό σημείο η συμφωνία του Μερκοσούρ θα μπορέσει να εγγυηθεί δισεκατομμύρια, πραγματικά δισεκατομμύρια επιπλέον εξαγωγών για πολλούς από τις τομείς μας, ακόμα και για τη Γεωργία παντού. Αναφερθήκατε σε κάποιους υποτομείς, για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, τα ωφέλη θα είναι τεράστια. Και οι θέσεις επίσης εργασίας θα είναι πάρα πολλές. Και επιπλέον μια τέτοια συμφωνία, ας τη δούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ζούμε σε έναν κόσμο που κάποιοι λένε ότι οι κανόνες δεν ισχύουν πια. Ποιος ενδιαφέρεται για τον ΠΟΕ, ποιος ενδιαφέρεται για τους διεθνείς κανόνες και το σεβασμό των κανόνων. Η συμφωνία του Μερκοσούρ είναι το τέλειο παράδειγμα στην καταλληλότερη χρονική στιγμή να δείξει ε, σε όλους αυτούς που εξετάζουν αυτό το λανθασμένο και προκατελημένο τρόπο ότι η μόνη λύση είναι συμπεφωνημένοι κανόνες. Να μην χάσουμε λοιπόν μόνο αυτή την τεράστια οικονομική ευκαιρία αλλά και την πολιτική ευκαιρία τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Μπορώ να σας πω το εξής ένα στα δέκα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε είναι από την Περκοσούρ και τα περισσότερα από αυτά θα ρυθμιστούν βάσει ε, της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με το Μερκοσούρ. Ένα στα δέκα, λίγο λιγότερο από το ένα στα δέκα, ένα στα έντεκα, άντε να κάνουμε και τον υπολογισμό πιο σωστά. 38 στι 425, υπολογίστε τα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι υψή τη σημασία να υποστηρίξουμε του εργαζομένου μα, να άρουμε αυτού του φραγμού και να δημιουργήσουμε αυτέ τι επιπλέον ευκαιρίε. Παρεπιπτόντω, εάν δεν εξασφαλίσουμε πρόσβαση στο Μερκοσούρ τώρα, μαντέψτε ποιο ε, θα απολαύσει, αν θέλετε, αυτό το χώρο. Δεν θα είναι εμεί, είμαστε εμεί. Η εμπειρία μου με την Κίνα είναι ότι ε, η τεράστια πρόσβαση της Κίνας στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και μπορούμε να γίνουμε και μοχλό ε, για δημιουργίε θέσει εργασία στην Κίνα, αν θέλετε, αντί για δημιουργίε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πω άλλα. Σημειώνω το σχόλιο ότι θα πρέπει να αναφέρουμε τις διπλωματικές δράσεις της, ε, ε στην, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωβουλευτές. Έχετε εδώ και τον συνάδελφο, τον Chris Πέρες όταν πηγαίνει η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σε τρίτη χώρα, να έρθετε σε επαφή μαζί του, θα σας πούμε τα πιο πρόσφατα ε, στοιχεία για την πρόσβαση στις αγορές, ώστε να έχετε και ένα πλήρες οπλοστάσιο για να μπορέσετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μας. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το πιο σημαντικό. Και ε, στη συνέχεια θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω, απαντώντας σε μία ερώτηση, την οποία δεν ξέρω πού να την τοποθετήσω. Υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσία. Και όλα καλά και άγια, διότι ζούμε σε ένα κόσμο συνωμοσιών. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Το θέμα της Ινδονησίας και, το... και άλλων χωρών και πού βρισκόμαστε όσον αφορά το RED 2 και το φινικέλαιο είναι ότι οι Ινδονήσοι πραγματικά προβλέπουν ότι θα προσφύγουν στον ΠΟΕ εναντίον μας. Ε, έτσι όμως πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχουν κανόνες και ξεκινάει η συζήτηση μέσω αυτών των μηχανισμών. Αυτό που δεν μας αρέσει και τόσο είναι ότι η, Ινδονησία στέλνει και ε, ε, ενδείξεις ότι ίσως θα προσπαθήσει να πιέσει κάποιους τομείς μας, δημιουργώντας επιπλέον φραγμούς. Αυτό δεν είναι σωστό ε, και δεν λειτουργεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο ε, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Και φυσικά με τις Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να προσέχουμε. Ναι, υπήρχε συμφωνία με τον πρόεδρο Γιούγκερ και τον πρόεδρο Τραμπ να δούνε τα θέματα του εμπορίου για τη σόγια. Έχει υπάρξει πολύ σημαντική αύξηση εξαγωγών σόγιας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σχετίζεται με θέματα βιωσιμότητας όπως το Φιλικέλαιο. Πρέπει λοιπόν να τα βλέπουμε ξεχωριστά όσο γίνεται και δείτε λίγο πώς έχουν οι τιμές στην αγορά. Υπάρχει λιγότερη διαθεσιμότητα άλλων πηγών σόγιας και μείωση στις τιμές εξαγωγής της σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων δεδομένων και των προβλημάτων που υπάρχουν στην Κίνα για πρόσβαση στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι σαφώς και μία απάντηση βάση της αγοράς ο Μάτε μου γράφει κάτι, εγώ γερνάω, ξεχνάω ερωτήσει, ζητώ συγγνώμη. Πώ ακριβώ ε, ε, φροντίζουμε να κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Είναι μια ερώτηση που μου διέφυγε, δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάποια άλλη, όχι γνέφει ο Μάτε. Η σύντομη απάντηση είναι μιλήστε με τον κύριο Λαντσίνη. Αυτό που έκανε ήταν ότι στη Λομβαρδία προετοιμάστηκε με πολλές τομιακές ενώσεις ε, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως και ξεκίνησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση που ήταν λιγότερο πολιτική φύσεω, αυτά που είστε συνηθισμένοι δηλαδή, αλλά ήταν πολύ χρήσιμη γιατί καταφέραμε να συμμετέχουμε κι εμεί. Δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε συνεχώ σε τέτοιε εκδηλώσει. Συμμετείχαμε όμω και παρουσιάσαμε τι υπηρεσίε που διαθέτουμε για τι επιχειρήσει μα. Και αυτό το εκτίμησαν ιδιαίτερω σε μια περιοχή όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυθονούν και φυσικά δεν είναι ε, τόσο ρευστά τα πράγματα όσο θα, θα έλαμε, γιατί δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Νομίζω ότι μπορεί να σας δώσω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και αν μας το επιτρέπει ο χρόνος θα μπορέσουμε εμείς να υποστηρίξουμε ε, τις προσπάθειές σας. Ε, σκεφτείτε όμως ότι ε, τι θα ήταν καλύτερο για να προσφέρετε αυτές τις πληροφορίες στις περιφερειές σας. Όταν το αποφασίσετε μιλήστε μαζί μας, με ξέρετε. Ο ΜΕΤΕ είναι το δεύτερο θύμα και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε με βάση και τους πόρους μας για να μπορέσουμε να δούμε με πώς με τον καλύτερο τρόπο θα προωθήσουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, στις κάτω χώρες, ε, στις ημέρες ε, της αγοράς ε, και αυτό που κάναμε στη Χάγη, είχαμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έγινε στην Κοπενχάγη πριν από μερικούς μήνες, διότι το ενδιαφέρον στα θέματα, στις παρουσιάσεις, στα εργαλεία που προτιμούν οι Ολλανδικές επιχειρήσεις και ενώσεις είναι διαφορετικό από αυτά που προτιμούν οι επιχειρήσεις στην Κοπενχάγη. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε λοιπόν όσο καλύτερο μπορούμε και να κάνουμε πράγματα στα μέτρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο 10 και περνάμε αμέσως στο σημείο 11. Μία σύντομη παρουσίαση των ε, σχετικών με τον εμπόριο πτυχών της Συνόδου G20 στην Οσάκα. Στις 28 και 29 Ιουνίου υπό η Ιαπωνική Προεδρία. Έχετε το λόγο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να τελειώσω εντός 5 λεπτά έχουν περάσει δύο μήνες από τη Σύνοδο και έχουμε ενημερωθεί για τη Σύνοδο των G7. Και στις δύο συνόδους το εμπόριο ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης, καθώς και οι καταχρήσεις ε, που, και παραβιάσεις που σημειώνονται από διάφορες χώρες υπήρξε μια συμφωνία για έναν μηχανισμό προστασίας ε, των ε, πολυμερών εμπορικών σχέσεων και επίσης υπήρξε συμφωνία για να δοθεί ένα κοινό μήνυμα. Βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο Χάλιβας απασχόλησε πάρα πολύ το G20 και το G7 και υπήρξε μια ε, συμφωνία γι' αυτό. Τώρα, οι πτυχές σχετικά με το εμπόριο της ε, Συνόδου Κορυφής στην Οσάκα είναι οι εξή ε, Το γενικότερο αφήγημα του εμπορίου γενικότερα, έπειτα το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ε, Χωρτικότητα χάλιβα και αυτό που έθεσε ως προτεραιότητα η Ιαπωνική Προεδρία είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο κυρωές δεδομένων. Αν προσπαθήσω να συνοψίσω το αποτέλεσμα της ε, συνόδου, θα μπορούσα να πω ότι από την οικονομική πλευρά ο Φρανσίσκος σας έδωσε μια εικόνα του που βρισκόμαστε. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν διάφορες εντάσεις στο εμπόριο οι οποίες κλιμακώνονται τους τελευταίους μήνες με ε, δασμούς ε, εκατέρωθεν από πολύ σημαντικούς παίκτε ε, στο παγκόσμιο εμπόριο. Τώρα, από πλευράς ε, διεθνούς διακυβέρνησης υπήρξε δυσκολία στην έβρεση συνένεσης στα σημαντικά εμπορικά ζητήματα. Δεν θα υπερβάλλω αν πω ότι ήταν σχεδόν αδύνατον να γίνει κάτι τέτοιο στις δύο τελευταίες υπουργικέ συνόδους του ΟΣΑ. Ε, στον ΟΣΑ δεν καταφέραν να συμφωνήσουν τα τελευταία τρία χρόνια οι συμφωνίε μάλιστα στις οποίες οδηγούνται είναι για δευτερεύουσα σημασία πράγματα. Και στην ε, G20 πέρυσι στον Buenos υπήρξε μια συμφωνία για την αναγκαία μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο, η σύνοδος στην Οσάκα ήρθε μετά από μια υπουργική ε, σύνοδο η οποία κατέληξε σε μια σημαντική ε, δήλωση που ναι μεν έδειξε τα ισχυρά σημεία αλλά και τα αδύναμα όπως η έλλειψη συνένεσης. Επαναλήφθηκε λοιπόν το μήνυμα της ανάγκης για μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και η αναγνώριση να αντι... του ότι υπάρχουν ε, προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο διεθνές εμπόριο. Σχετικά ενημέρωσα και τους ε, συναδέλφους σας πρόσφατα. Επίσης χρειάζεται και μία νέα αντιμετώπιση της ε, νομοθεσίας ώστε να γίνουν αλλαγές. Μετά συζητήθηκε το, συζητήθηκαν, συζητήθηκαν οι στρεβλώσεις στην αγορά και οι πιέσεις που ασκούν και το θέμα των επιδοτήσεων. Φυσικά υπήρχε διαφωνία μεταξύ των ηγετών. Συζητήθηκε επίσης και το ζήτημα του πλεονάσματος χάλιβα στο μέλλον. Ούτε και εδώ βρέθηκε συνένεση. Κυρίως για λόγους που αφορούσαν την ουσία και δευτερευόντως για διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Έπειτα, η έκθεση για τις ε, δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΠΟΕ συζητήθηκε, συζητήθηκαν τα επιτυχίες που αφορούν την ε, διαφάνεια και τις διεθνείς δεσμεύσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αναγνωρίστηκε ε, το πόσο σημαντικό είναι να αναλυφθεί δράση. Επίσης, η έκθεση που λάβαμε από την ε, Γενική Γραμματεία και από την Προεδρία αναφέρει ότι ήταν από τις ε, πιο δύσκολες συνόδους G20. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην δημοσίευση μιας κοινή δήλωσης υπήρχε δυσκολία συνεννόηση τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και σε επίπεδο υπουργών για μια κοινή θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είχε εξέχοντα ρόλο. Ο πρόεδρος Γιούνκερ απίφθινε ένα κτίριο λόγο μετά τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας τόνισε τη σημασία του διεθνούς εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύνοδο ήταν να προσπαθήσει να βρεθεί συνένεση για τα δύσκολα ζητήματα και για παράδειγμα για την διαχείριση των διεθνών εντάσεων. Καταφέραμε όμως οι γενικές γραμμές να ακολουθήσουμε τις ε, γραμμές μας. Ε, θα καλωσορίσουμε την κοινή δήλωση των Υπουργών και το κείμενο στο οποίο θα συμφωνήσουν. Στο κείμενο αυτό θα γίνεται αναφορά στο ελεύθερο εμπόριο, στις ανοιχτές αγορές, στη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και σε αλλαγή συμπεριφοράς έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του. Αναφορά θα γίνεται επίσης στο ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω τα πέντε λεπτά, αλλά θα αναφερθώ σύντομα στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την, ε, το Παγκόσμιο Πλεόνασμα Χάλιβα. Στην Σύνοδο ακούστηκε ότι πρέπει να συνεχίσει η λειτουργία του φόρουμ αυτού έτσι ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ε, κρατών. Βέβαια, οι ηγέτες ε, συμφώνησαν ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να επιστρέψει στα χέρια των αρμόδιων υπουργών και το φθινόπωρο φέτος, το 2019, θα συζητηθεί ξανά. Μετά την ε, Σύνοδο δημοσιεύτηκε και μία κοινή δήλωση, συνυπογεγραμμένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη δήλωση όμως δεν συμμετείχαν τρεις σημαντικές χώρες. Ινδονησία, Νότια Αφρική. Και στη δήλωση αυτή συμφωνήθηκε να δοθεί όθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τόνωση στο εμπόριο γενικότερα αυτό που συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση τριμερώς με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ιαπωνία είναι να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στο διεθνές εμπόριο. Αυτά προς το παρόν. Με χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο, εκτός από το Χέλμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Ένα σύντομο σχόλιο γιατί αναφέρατε το φόρουμ και τη θέση που βρισκόμαστε. Ποια θέση έχει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, τη συνέχιση του φόρουμ CST. Uh, Ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε μια πιο σαφή αξιολόγηση και να μας περιγράψετε τι συνέβη ακριβώς εκεί. Αν δεν απατώμε, λέτε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο, δεν βλέπει τίποτα ούτε για το φόρουμ του, του Χάλιβα, ούτε για την ε, μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Πώς το βλέπετε και πώς ε, έτσι περιμένετε να έχει το μέλλον είναι δαπανηρό αυτό το εγχείρημα και δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθειες σε σχέση με την παρούσα κατάσταση ή έχει νόημα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Για το φόρουμ για το Χάλιβα, νομίζω ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και η θέση ε, των 19, των 18 από το G20, είναι σαφέστατα να επιμείνουμε στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί στις υπουργικές διασκέψεις των Παρισίων και του Βερολίνου για την μείωση της υπερβολικής δυνατότητας και παραγωγής ε, και των συμπαραματούν των ε, φραγμών στο εμπόριο και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό μέχρι ε, τη Σύνοδο Κορυφής των G20 υπό Κινέζικη Προεδρία που είναι προθεσμία να παραταθεί τότε η εντολή του Παγκοσμίου Φόρουμ. Είναι σχεδόν ομόφωνη η επιθυμία στο G20 να παραταθεί. Τώρα θα πρέπει να φέρουμε στο πλευρό μας τον έναν ή τους δύο που ακόμα διαφωνούν από τους G20. Βέβαια αυτό είναι πολιτικό εγχείρημα και δύσκολες οι συνθήκες. Η του δυο που ακομα διαφωνουν απο του g 20 λέγει εγχειρημα και δυσκολε οι ήταν λογικό το αποτέλεσμα έτσι, σόφρων δεδομένων και των συνθήκων και των διεθνών σεναρίων στο εμπόριο. όπου έχει έρθει ένας κατακλυσμός και εφαρμόζονται μέτρα, επιβάλλονται μάλιστα εκτός του πλαισίου του ΠΟΕ. Το γεγονό ότι ακόμα υπάρχει συζήτηση και κάπου μπορεί να διαγραφεί μια βασική συνένεση για κρίσιμα θέματα, όπως είναι η ανάγκη ε, φερρυπίν ε, διατήρηση και βελτίωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το G20 και το G7 θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι φόρουμ διαπραγμάτευσης, είναι ε, φόρα συζήτησης, παγκόσμιας διακυβέρνησης, ανταλλαγής απόψεων, αλλά δεν παίρνουν αποφάσεις, πόσο μάλλον για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Είναι σημαντικό να συζητούν ε, οι ηγέτες τα σημαντικά και να προσπαθούν να σφυριλατούν κάποια συνένεση. Για τις μεταρρυθμίσεις όμως, στον ΠΟΕ, αυτό είναι άλλο θέμα. <laughs> Χθες είχαμε μια πρώτη γεύση έτσι, ε, σχετικά με τα όσα θα συζητηθούν στον ΠΟΕ που είναι ακόμα σε θερινές διακοπέ και θα συνεχιστούν οι συνομιλίες την άλλη εβδομάδα. Πάντως χρειάζεται πολιτική στήριξη από το G7 και το G20. Προς το παρόν εκεί βρισκόμαστε. Στον όσα. που είναι και ομονοούσε οι χώρε, δεν υπήρξε δήλωση ε, επί μια τριετία, πόσο μάλλον εκεί που διαφωνούν οι χώρες. Υπάρχουν ε, μεγάλες ε, διαφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων πρωταγωνιστών και δεν το κρύβουμε άλλωστε, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό. Αλλά μπορούν οι g να συμφωνήσουν για κάποιους κανόνες, είδους κανόνες παιχνιδιού, ελεύθερο εμπόριο, δίκαιο. Του χρόνου ε, ε, θα γίνει υπουργική διάσκεψη για τον ΠΟΕ. Γενικά ε, το G20 και το G7 μπορεί να στείλει ένα θετικό μήνυμα, ένα θετικό πνεύμα. Οι δράσεις θα ακολουθήσουν όπου πρέπει να ληφθούν αυτές, να αναλυφθούν είτε μονομερός είτε διμερός. Α, προηγουμένως ξέχασα να αναφέρω την ανακοίνωση Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του G20 στο BRH και το δέχτηκαν πάρα πολύ θετικά στο G20 στην Οσάκα, για να υπάρξουν λύσεις που να βασίζονται σε κανόνες στο εμπόριο υπό δύσκολες συνθήκες. Εκεί βρισκόμαστε. In Προ τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Εύκολο δεν είναι το εγχείρημα γιατί δίστανται, όπω είπαμε, οι απόψει για τα διάφορα θέματα. Από τη μια έχουμε προστατευτισμό, από την άλλη επενδυτικές ε, ε, ε, ενισχύσει και στρεβλώσεις τη αγορά. Πάντω όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κέντρο τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά πάντα είναι καλύτερο να συζητάς παρά να μην συζητά με τον άλλον. Ε, και για μια ελπίδα ζούμε ως γνωστόν. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ολοκληρώνεται το σημείο 11 εδώ και προχωρούμε στο 12 που είναι η επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για το εμπόριο μεν, αλλά και για τις επενδύσεις εκτός από το εμπόριο και τα τελευταία χρόνια είχαν ε, γίνει σκληρές συζητήσεις ε, για το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, για τη μεταρρύθμιση αυτού του συστήματος και για τις συζητήσεις γενικότερα στα πλαίσια του ΠΟΕ σχετικά με τη ε, διευκόλυνση των επενδύσεων. Πολλά λοιπόν τα τεκτενόμενα και τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε πού βρισκόμαστε και χαίρομαι πολύ που έχω δύο βασικούς εμπειρογνώμονες εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα επενδύσεων. Έχουμε τον Κάρλο Πετινάτσο και τον Κόλιν Βόρμ δίπλα του, που είναι οι εμπειρογνώμονες για θέματα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε κάποια σχόλια για τις πρόσφατες ε, εξελίξεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον ΠΟΕ, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος διευθέτης διαφορών επενδυτή κράτους και το Διεθνές Επενδυτικό Δικαστήριο. Και εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συζητάμε αυτά. Και υπάρχει και το θέμα της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Χάρτη θα θυμάστε ότι είναι η μόνη συνθήκη που έχει κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το παλιό σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους και πολλά θέματα έχουν να κάνουν με την ενέργεια, ακόμα και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, πόσο μάλλον με τους επενδυτές. Άρα απαιτείται επιγόντως ε, μεταρρύθμιση. Νομίζω θα αργήσει ο Κάρλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι εδώ στην Επιτροπή. Είναι η πρώτη μου παρέμβαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική εισαγωγή. Θα ήθελα εν συντομία να σας ενημερώσω για τέσσερα σημεία στις διαπραγματεύσεις μας ε, στο θεματολόγιο μας και ε, φυσικά ο συνάδελφος θα ολοκληρώσει με το θέμα της επίλυσης διαφορών και της ε, πολυμερής ε, εξελίξης. Τα τέσσερα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ εν συντομία είναι οι πιο σημαντικές διαπραγματεύσεις, οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τις επενδύσεις, η διαδικασία διευκόλυνσης των επενδύσεων του ΠΑΟΕ, η συνθήκη της ενεργειακής χάρτας, εξυγχρονισμός της συνθήκης και δύο λόγια για το screening και για το τι κάνουμε για να εφαρμόσουμε ε, το νέο εργαλείο screening ε, των ξένων επενδύσεων, του ελέγχου ουσιαστικά των επενδύσεων. Όσον αφορά την Κίνα, ε, αυτή θα είναι η πρώτη ε, ξεχωριστή συμφωνία επενδύσεων, προστασίας των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πλήρη ε, συμφωνία γιατί καλύπτει και την προστασία και την απελευθέρωση. Γι' αυτό ακριβώς και την αποκαλούμε συνολική συμφωνία. Θα αντικαταστήσει ταυτόχρονα, αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ, τις 26 κείμενες ε, διμερείς συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων που έχουν ήδη τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για παλιότερες φυσικά συμφωνίες. Ο βασικός στόχος για μας είναι να δώσουμε μια νέα ισορροπία στο επίπεδο πρόσβασης και στις συνθήκες για να επενδύσουν οι επιχειρήσεις μας στην Κίνα και να δώσουμε μια νέα ισορροπία γιατί φυσικά η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις πιο ανοιχτές και ευνοϊκέ στον κόσμο και θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο ε, επίπεδο ισον, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην Κίνα. Αυτό είναι ο στόχος. Η δήλωση της Συνόδου φέτος ήταν πάρα πολύ σημαντική διότι συμφωνήσαμε ε, εκατέρωθεν να βελτιώσουμε ουσιαστικά την πρόσβαση στις αγορές και τις συνθήκες την άρση ε, διακριτικών απαιτήσεων και πρακτικών που παρακολούν τους επενδυτές και ε, τη δημιουργία ενός ισορροπημένου πλαισίου προστασίας επενδύσεων που περιλαμβάνει και όρους για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επόμενος γύρος θα είναι αυτό το μήνα στο Πεκίνο την εβδομάδα της 23ης Σεπτεμβρίου και συμφωνήσαμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα κάνουμε έναν απολογισμό και θέλουμε να σταθούμε κυρίως στη βελτίωση των προσφορών μας, ε, των προσφορών πρόσβασης της αγοράς. Έχουν γίνει ήδη ανταλλαγές προσφορών και ο στόχος φέτος είναι να γίνει ουσιαστικό πρόεδρος ε, για αυτές τις προσφορές για την πρόσβαση στις αγορές. Ο τελικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία το 2020. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτό ε, δεσμεύτηκαν να κάνουμε δύο πλευρές. Αυτά για την Κίνα. Δεύτερο, διευκόλυνση επενδύσεων του ΠΟΕ πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία. Είναι η λεγόμενη κοινή υπουργική πρωτοβουλία που σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει όλα τα μέλη του ΠΟΕ είναι σαν μια πολυμερή πρωτοβουλία μιας ομάδας ε, περίπου 70 μελών με στόχο να συμφωνήσουμε τελικά σε ένα πολυμερές πλαίσιο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων που θα καλύπτει όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση. Ε, ξεκίνησε από μια ομάδα αναδυόμενων χωρών, δεν προτίθηκε αρχικώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αναπτυσσμένε χώρε, αλλά κυρίω από τη Λατινική Αμερική, την Κίνα και άλλου αναδυόμενες χώρες. Εμείς ε, ε, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή τη δήλωση και δεσμευθήκαμε και ενεργά στις ε, ε συζητήσεις στη Γενέβη και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει υπάρξει καλή πρόοδος, ότι οι συζητήσεις οδεύουν προς σχεδόν ένα στάδιο διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα στο δεύτερο εξάμεινο, γιατί πλέον συζητούμε για πιθανές διατάξεις μιας πολυμερούς συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Τι είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, δεν είναι η πρόσβαση, ε, ούτε η προστασία των επενδύσεων, είναι το ισοδύναμο μιας συμφωνίας διευκόλυνσης εμπορίου. Δηλαδή, να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες επενδύσεων, το επίπεδο διαφάνειας, τα διοικητικά, το διοικητικό άχθος που πολλοί επενδυτές μας λένε ότι ορισμένες φορές είναι και η ουσία του προβλήματος. Τα βασικά προβλήματα για επένδυση σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες ακριβώς, πού να βρούνε τι, ε, και το διοικητικό άχθος είναι τεράστιο. Γι' αυτό ακριβώς ε, και θεωρούνται ότι είναι τα βασικά προβλήματα ε, και οι βασικές ανησυχίες για ξένες επενδύσεις. Υπάρχει κάτι σημαντικό λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία και από συστημική σκοπιά, διότι θα ε, δείξει το δυναμισμό του ΠΟΕ, εάν προχωρήσει όντως αυτό ως πρωτοβουλία, η οποία στη συνέχεια θα γίνει ένα πολυμερές πλαίσιο. όσοι έκαναν την πρόταση, αλλά και ο Γενικό Διευθυντή, ο Χεσεβέδο, είπε ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε κάποια παραδοτέα στην επόμενη υπουργική διάσκεψη που θα γίνει του χρόνου. Ίσως λοιπόν αυτό να σημαίνει κάτι, μάλλον όχι τελική συμφωνία, αλλά θα έχει γίνει ουσιαστικό πρόεδρος, ε, πρόοδος για τη δημιουργία αυτής της ε, νέας ε, συμφωνίας. Υπάρχει εντολή στο Συμβούλιο ήδη και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει την εντολή πριν το τέλος του μηνός για να είμαστε και έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με όλους τους υπολείπους. Τρίτον, εξυγχρονισμό ε, τη συνθήκη ενεργειακή χάρτα. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Όλα τα μέλη της ενεργειακής χάρτας έχουν συμφωνήσει να γίνει ο εξυγχρονισμός των διατάξεων. Πρόκειται για κάτι το οποίο συντάχθηκε στη δεκαετία του 90. Δεν ανταποκρίνεται λοιπόν πλέον ε, στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προστασία της ενέργειας και η συμφωνία αυτή, όπως είπατε, δημιουργεί πολλές ε, διαφωνίες και οι διαφωνίες βασίζονται σε κανόνες οι οποίοι δεν είναι τόσο σαφώς καθορισμένοι όσο είναι πλέον οι κανόνες προστασίας των επενδύσεων στις σύγχρονες συμφωνίες μας. Δεν υπάρχει, ε, όπως είπε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, σαφές δικαίωμα να ε, ρυθμίσουμε τα πράγματα, ενώ όπως είπε το δικαστήριο θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξυγχρονιστεί αυτή η συμφωνία και να μπορέσουμε να την ευθυγραμμίσουμε στο σύγχρονο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους κανόνες προστασίας των επενδύσεων ε, οι διαπραγματεύσεις κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουν αρχές του 2020. Βρισκόμαστε σε μια φάση προδιαπραγμάτευσης, αν θέλετε, όπου η κάθε πλευρά καθορίζει τους στόχους τους. Δεν θα είναι εύκολο φυσικά, δεν είμαστε τα μόνα συμβαλόμενα μέρη, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρόκειται για μια περιφερειακή συμφωνία πολυμερή και θα δούμε. Μεγάλη πρόκληση, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για μας. Τέλος. Δύο λόγια για το screening των ξένων επενδύσεων. Φέτος ε, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα κράτη-μέλη έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ για την προετοιμασία της ε, εφαρμογής η οποία θα ξεκινήσει, ο μηχανισμός συνεργασίας δηλαδή θα ξεκινήσει ε, τον Οκτώβριο του 2020. Ο κανονισμός ήδη ισχύει, αλλά αυτό το σκέλος, η συνεργασία που είναι και η ουσία του μηχανισμού θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 και έχουμε αρχίσει να ε, προετοιμάζουμε όλη την εργασία και το μηχανισμό συντονισμού εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη, ε, δημιουργώντας όχι μόνο τον ασφαλή διάβλο επικοινωνίας που πρέπει να συσταθεί εκ νέου, ε, διότι πρόκειται για πολύ εμπιστευτικά δεδομένα και πληροφορίες και η ανταλλαγή τους ε, πρέπει να γίνεται με πολύ εμπιστευτικό τρόπο, γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διάβλος, πρέπει να συστηθεί ένας καινούριο και ε, πρέπει να καθορίσουμε όλες τις διαδικασίες εσωτερικά, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει γνωμοδότηση για όλες τις συναλλαγές, για ξένες επενδύσεις, σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες ασφάλειας ή δημοσίας τάξεως και ε, η γνωμοδότηση, η γνώμη θα πρέπει να διαμορφώνεται εντός 35 ημερών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυση και μετά να γνωμοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των συναλλαγών και θα υπάρχουν φυσικά πάρα πολλές συναλλαγές, διότι η Ευρώπη ε, λαμβάνει πολλές ε, ξένες επενδύσεις. Προπαρασκευαστικά λοιπόν μεγάλη πρόκληση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιστρέψουμε εδώ στην Επιτροπή και ε, δεν θα έχουμε μία ε, συνοπτική ε, εξήγηση ε, που είναι αυτό που εξηγεί συνοπτικά τι έχει γίνει από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός στις αρχές του έτους και όλα τα στάδια μέσω της ε, διαπραγμάτευση θα έρθουμε να σας τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τέλος για το screening έχουμε ε, και πολύ καλή συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την ε, Ιαπωνία σε τριμερές πλαίσιο, γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο, δεδομένου ότι είναι πολύ καλή η εμπειρία που διαθέτουν ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία εδώ και χρόνια στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κάλλο για αυτήν την ε, περιεκτική παρουσίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ε, πολυμερή μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης επενδυτικών διαφορών ιδιαίτερα για το Πολυμερές Επενδυτικό Δικαστήριο. Έπειτα, για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών και για την ε, Σύμβαση του Μαυρίκιου, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία ε, εδώ και αρκετό καιρό. Όπως είπατε λοιπόν και εσείς κύριε Λάγκε, Όλα αυτά η Επιτροπή τα στήριζε και στο παρελθόν. Τώρα έχει λάβει την έγκριση από το Συμβούλιο το Μάρτιο του 2018 για να διαπραγματευτεί ε, πάνω στο Διεθνές Πολυμερές Δικαστήριο. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Η συζήτηση για την ενδεχόμενη δημιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου γίνεται σε επίπεδο ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της ε, ομάδας εργασίας για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Είναι η ομάδα 3 που εξετάζει την ε, δεχόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών. Είναι ανοιχτή η ομάδα εργασίας υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Την, ε, στην τελευταία συνεδρίαση συμμετείχαν 106 χώρες. Όλα τα έγγραφα είναι στην ε, ιστοσελίδα της ε, Κομισιόν. Υπάρχουν γραπτές εκθέσεις, οι οποίες είναι επίσης ε, διαθέσιμες και δημοσιεύονται λίγο μετά το, την εκάστοτε συνεδρίαση. Υπάρχει οπτικο-ακουστικό υλικό σε όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών. Να τονίσω επίσης τα εξής, ότι υπάρχει ένα ταμείο το, στο οποίο συνεισφέρουν αρκετές ε, χώρες ε, προς τα ταξιδιωτικά έξοδα αναπτυσσόμενων, ε, εκπροσώπων από αναπτυσσόμενες χώρες έτσι, ώστε να μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις συνεδριάσεις. Έγιναν λοιπόν αρκετές συνεδριάσεις ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2017 και πλέον έχει συμφωνηθεί ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα σε ό,τι αφορά το σύστημα επίλυσης διαφορών. Απέχουμε πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα πρέπει να γίνουν βήματα έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην έγκριση μιας νέας συμφωνίας. Τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένες ε, οι επόμενες συνεδριάσεις στη Βιέννη, τον Απρίλιο του 2020 στη Νέα Υόρκη και έχουμε συμφωνήσει ότι θα αφιερώσουμε χρόνο για να εξετάσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στο πλαίσιο της ε, σύστασης αυτού του Διεθνούς Δικαστηρίου επενδυτικού δικαστηρίου. Μεταξύ δύο συνεδριάσεων γίνεται και μία ενδιάμεση ε, συνεδρίαση. η οποία συνδέει τις ε, δύο κύριες ε, συνεδριάσεις. Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις ενδιάμεσες συναντήσεις είναι να παρουσιαστεί το έργο που έχει ήδη γίνει και να, παρουσιαστούν, να παρουσιαστούν οι απόψεις των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδιαίτερα των χωρών ε, της Αφρικής και των ε, γαλλόφωνων συγκεκριμένα χωρών της Αφρικής. Η συνολική μας εκτίμηση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Όπως σας είπα, στην τελευταία συνάντηση ήταν παρούσε σε 106 χώρες. Υπάρχει γενικότερα συνένεση για να γίνουν ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στην ιστοσελίδα σχετικά με αυτό θα βρείτε τις ε, σχετικές πληροφορίες καθώς και τις προτάσεις που έχουν γίνει. τον Ιανουάριο του 2019 δημοσιεύσαμε τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές ε, για το ποια θα πρέπει να είναι η δομή του Διεθνούς Επενδυτικού Δικαστηρίου. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό θα προχωρήσουμε, θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές, προτού περάσουμε ε, στο, σχέδιο του, στο στάδιο του σχεδιασμού. Αυτό θα πάρει περίπου δύο χρόνια. Επίσης, ήθελα να σταθώ λίγο στο έξι, στο Κέντρο Επίλυσης Διαφορών, το οποίο ασχολείται με την επίλυση επενδυτικών διαφορών. Το κέντρο αυτό αποφάσισε να επικαιροποιήσει τους κανόνες λειτουργίας του, χωρίς όμως να γίνει κάποια αλλαγή στη σχετική συνθήκη σύστασής του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκεται υπό επεξεργασία η τρίτη βεσιόν των κανόνων λειτουργίας του κέντρου αυτού. Η επόμενη συνάντηση για το σκοπό αυτό θα γίνει το Νοέμβριο. Τα κράτη-μέλη πιέζουν για να γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη συμφωνηθεί διμερώς. Όπως σας είπα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά συζητούμε θέματα διαφάνειας, χρηματοδότησης των τρίτων μερών και ε, θέματα που αφορούν ε, κανόνες σχετικά με το αν θα είναι παραδεκτή ή όχι μία προσφυγή. Περιμένουμε λοιπόν αποφάσεις στις αρχές του επόμενου έτους που θα εξαρτηθούν από την συνάντηση του Νοεμβρίου. Τέλος, η σύμβαση του Μαυρίκιου. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι αφορά την διαφάνεια στο σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή ε, και κράτους. Προβλέπονται λοιπόν διάφορες παρεμβάσεις χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες και το σκεπτικό είναι οι κανόνες αυτοί να εφαρμοστούν στις υφιστάμενες ε, συνθήκες για, για την επίλυση επενδυτικών διαφορών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως υπόδειγμα για την σύσταση του επενδυτικού δικαστηρίου. Ο κύριος Λάγκε και η Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από το Συμβούλιο του 2015 να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ο φάκελος αυτός είχε κάποιες καθυστερήσεις, όμως φέτος συζητήθηκε εκ νέου στο Συμβούλιο, το οποίο αναγνωρίζει ότι για να μπορέσει να προβεί σε αλλαγές θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Έχουμε μία μικρή μειοψηφία κρατών μελών που αρνούνται να υπογράψουν τη σύμβαση αυτή. Όπου, όπως σας είπα, είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν στο Συμβούλιο να πιέσουμε έτσι ώστε να εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Αυτά λοιπόν από μένα προς το παρόν. Ευχαρίστω θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας και όπως είπε ο Κάρλο θα ξανάρθουμε στην Επιτροπή σας και θα ερχόμαστε συχνά για να σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σένα. Κόλιν. Κόλιν, Μπορείς να κατονομάσεις, σε παρακαλώ, τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση του Μαυρικίου και δεν είναι υπέρ της δυναφάνειας και στη διαδικασία επίλυσης διαφορών επενδυτή Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κατονομάσω τις χώρες αυτές, αλλά οι χώρες που είχαν τα περισσότερα προβλήματα, γενικότερα με τη διαφάνεια, και που έχουν και θέματα με το κράτος δικαίου. Πώς να το πω, να το πω αλλιώς. Το σημαντικότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχει διαφάνεια ο ενεργειακός χάρτης. Δηλαδή βασικά τα Υπουργεία Ενέργειας είχαν κάποια ζητήματα και δυσκολίες. Ελπίζω τώρα να καταλάβατε ποιον ε, κρατών πρόκειται. Πας για το διπλωματικό σώμα. Πολύ διπλωματικά μας τα λες. Η Μακουλάδα Ροτρίγκες Πινέρο. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εκπροσώπους ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή τους. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο κύριος Πεκινάτου μας είπε στην αρχή και συμφωνώ μαζί του ότι είναι σημαντικές οι πολιτικές των επενδύσεων ε, ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα δεσμευτικό σύμφωνο και να συνδέονται οι επιχειρήσεις και επενδύσει με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα όμω δεν έχουμε στο Συμβούλιο, ε, δεν μας έχει δώσει ε, την εντολή. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποκτήσει εντολή από το Συμβούλιο για να γίνει κανονική διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά το πολυμερέ ε, διεθνές επενδυτικό δικαστήριο. Ποιος και με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει τη συνέχεια και συνέπεια των αποφάσεων των διαιτητικών που μπορεί να αποκλείουν μεταξύ τους. Θα υπάρξει νομολογία, όπως υπάρχει στα τακτικά δικαστήρια και σε ένα τέτοιο διαιτητικό όργανο και πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. επίσης θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Πώς προβλέπετε να ε, καταλήγετε και πότε σε αντίστοιχη συμφωνία. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω 106 χώρες εργάζονται σε αυτό το θέμα. Συμμετέχει εκεί η Ιαπωνία. Και ποια είναι η στάση της ε, ως προς τη διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία των Επενδύσεων που συζητάτε εκεί. Και τέλος, για τις διαπραγματεύσεις ε, με την Κίνα. Τι γίνεται με το δρόμο του μεταξιού. και μπορεί να μπει και η δική μας θέση για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ως προς αυτό το σχέδιο του δρόμου του μεταξύ που έχει κάνει η Κίνα. Ευχαριστώ. Ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη λεπτομερή παρουσίαση ε, της κατάστασης από τους δύο ε, εμπειρογνώμονες. Έχω και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, για τον ενεργειακό χάρτη. Περιγράψατε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και τον επόμενο γύρο στις αρχές του επόμενου έτους. Κάποιες χώρες, μέλη, αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τον ενεργειακό χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει το παράδειγμα κάποιων κρατών μελών που αποχωρούν από τον ενεργειακό χάρτη. Γιατί αν δεν προχωρήσει τα μεταρρύθμιση, όπως είπατε, είναι πιο εύκολο να φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ενεργειακό χάρτη. Δεύτερη ερώτηση προς τον Κόλιν. Ξέρουμε αυτά τα θέματα τα επενδυτικά και με το διαιτητικό διεθνές έτσι, πολυμερές δικαστήριο. Υπάρχει τώρα όμως κανένα μήνυμα ή κανένα σημάδι ότι αυτό δεν αφορά μόνο την άμεση προστασία των δικαιωμάτων ε, των επενδυτών, αλλά ένα τέτοιο διεθνές διαιτητικό δικαστήριο θα ασχοληθεί και με τις υποχρεώσεις των επενδυτών, εγχώριων και αλλοδαπών. Γιατί υπάρχουν τα δικαιώματα των επενδυτών, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις τους. Μπορείτε λοιπόν να μας απαντήσετε. Δηλαδή θα λειτουργεί ως ένα κανονικό δικαστήριο ως άοφιλε. Η κυρία Μπρινκμό. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας ε, για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς τη συμβατότητα ε, με τις ευρωπαϊκές συνθήκες του Δικαστηρίου Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους. Ε, δεν σας κρύβω ότι δεν ε, έχουν ξεπεραστεί οι φόβοι μας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπήρξε η απόφαση το 2017, αλλά ξέρουμε ότι οι διάφορες επιχειρήσεις ε, πετρελαϊκές ε, κάνουν πολλές έρευνες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Ε, και για να φτάσουμε στους στόχους του Παρισίων, όλα τα αποθέματα και τα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να μείνουν στο υπέδαφος. Ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, επειδή θα υπάρξουν επιθέσεις και προσφυγές ε, από αυτό το κλάδο των πετρελαϊκών και των ανοιχτών καυσίμων, κινδυνεύουν να δικαιωθούν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κάνιας. Φαίνεται λίγο παράδοξο το εξής γεγονός. Ε, ε, ρωτάμε ποιε είναι οι χώρε αυτές που δεν θέλουν να υπογράψουν μια σύμβαση, τη σύμβαση του Μαυρικίου για τη διαφάνεια και εσεί μας απαντάτε ε, ότι δεν μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες αυτές. Μα πρόκειται για διαφάνεια, να τις κατονομάσετε, παρακαλώ. Επίσης, ακούσαμε ότι πρόκειται να συμφωνηθεί η θεωρητική βάση και η αντίληψη επάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το Διεθνές Διαιτητικό Πολυμερές Δικαστήριο. Δηλαδή ακόμα εκεί είμαστε στο στάδιο της σύλληψης και του σχεδιασμού του δικαστηρίου αυτού. Ρώτησε και είμαι Ροτρίγε Περέρο. σε ποιο χρονικό ορίζοντα κινούμαστε και μπορείτε να διακινδυνεύσετε κάποια πρόβλεψη. Να μας πείτε πότε περίπου σκέφτεστε ότι θα έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ και από πλευρά μου, λέει ο Πρόεδρος, εδώ και μια πενταετία βλέπω τον προγραμματισμό το χρονικό. Ε, πότε προβλέπετε κάθε ε, πράγμα να έρθει και πότε να λήξει. Και η περίφημη ρήτρα εκπνοής το 2020 η ε, ρήτρα grandfathering όπως λέγεται στα αγγλικά ε, για, το πότε θα λήξουν κάποια κεκτημένα παλαιά δικαιώματα του παρελθόντος. Υπάρχει ένας κανονισμός του 2012 ε, για τον εξυγχρονισμό του, των παλαιών τύπου συμφωνιών. Εμείς πότε όμως να περιμένουμε κάποια δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το τομέα. τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων. Εννοώ, Κάρλο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, προς τον ε, κύριο Ροντρίγκε Πινιέρο. Αναφέρθηκε στη θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δεσμευτική Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συζητήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Ισημερινού πριν από μερικά χρόνια και κάπου σταμάτησε, επιβραδύνθηκε και τώρα μόλις λάβαμε αναθεωρωμένη εκδοχή του κειμένου το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες. Δεν θα έπρεπε να πω για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτά είναι θέματα ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τα ε, συντονίζει και τα αντιμετωπίζει κατά βάση η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη-μέλη. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί ε, τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Να σας δώσω απλώς ε, μία εικόνα της κατάστασης. Δεν είναι και μυστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούσε κυρίως για τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διεξαγωγή της, αλλά και το πεδίο εφαρμογής ε, που είχε παρουσιαστεί αρχικώς ε, από όσους έκαναν την πρόταση. Το πεδίο εφαρμογή ε, ουσιαστικά κάλυπτε μόνο ξένες επιχειρήσεις. Προβλεπόταν λοιπόν υποχρεώσεις μόνο για ξένες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο είπαμε, για να το πω λίγο πιο απλά εδώ, ήταν ευθύ εξ αρχής ναι, ε, εμείς ε, πάντα υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με υποχρεώσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να μιλήσουμε για υποχρεώσεις για όλους. Κυβερνήσεις, ξένες επιχειρήσεις και εγχώριες επιχειρήσεις. Όλοι θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή ήταν η βασική μας θέση ευθύ εξ αρχής και Λάβαμε πάρα πολλές επικρίσεις ε, από αρκετούς, γιατί ίσως ήμασταν και οι μόνοι εκπρόσωποι του ανεπτυγμένου κόσμου που συμμετείχαν στις συζητήσεις, διότι όλοι οι υπόλοιποι αγρόνι γόραζαν, ούτε εμφανιζόντουσαν. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρούσα και τόνιζε τα θέματα αυτά και ελπίζω τουλάχιστον η συζήτηση τώρα να πάει προς μια πιο ισορροπημένη κατάσταση ε, έχουμε ένα νέο αναθεωρημένο κείμενο. Θα δούμε το πεδίο εφαρμογή και φυσικά θα ε, καταλήξουμε στη θέση μα με τα κράτη-μέλη και θα, σε μια προσπάθεια να είμαστε επικοδομητικοί. Δεν ε, θα προσπαθήσουμε σε καμία περίπτωση να παρακολύσουμε τη διαδικασία. Πρέπει όμω όλα να είναι ισορροπημένα και να περιλαμβάνουν τα πάντα. Δεν ξεχνάμε βεβαίως και τι ευθύνε των επενδυτών μας. Ε, αυτό το καλύπτουμε και στις ε, δικές μας τι συμφωνίε. Υπάρχουν ε, διατάξεις για την ευθύνη των επενδυτών. Ε, το αναμενόμενο είναι να συμπεριφέρονται σε κάθε τρίτη χώρα όπως κάνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δηλαδή διατάξεις από αυτού και στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά επίσης είναι σαφές ότι δεν μπορεί ο κάθε επενδυτή να χαίρει της προστασίας που προσπαθούμε να επιτύχουμε στις συμφωνίες μας, διότι ο επενδυτή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο βάσει και τη εγχώρια νομοθεσία. Εάν ένα ξένο επενδυτή δεν τηρεί του κανόνε τη χώρα στην οποία επενδύει, τότε δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την συγκεκριμένη προστασία. Αυτό είναι βασικός κανόνας. Η δεύτερη ερώτηση που θέσατε ήταν τι κάνουμε με την πρωτοβουλία για το δρόμο του μεταξιού ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Κίνα και τη Συνολική Συμφωνία για τις Επενδύσεις. Δεν ασχολούμαστε με την πρωτοβουλία αυτή, αυτή καθεαυτή. Ε, αυτό που ελπίζουμε είναι ότι θα μας βοηθήσει να εγγυθούμε τις συνθήκες για τους επενδυτές, όχι μόνο για τους επενδυτές μας στην Κίνα, αλλά σε αυτή την περίπτωση ε, σκεφτόμαστε και την διαφάνεια ε, των όσων χαίρουν κινέζικων επενδύσεων, διότι υπάρχουν και αρκετές ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό. Μέσω αυτή τη συμφωνίας προσπαθούμε να έχουμε το μέγιστο επίπεδο διαφάνειας και να υποστηρίξουμε το σεβασμό των διεθνών προτύπων. Και φυσικά πολλά από αυτά αφορούν τους κανόνες ε, ε, προμήθειών που δεν είναι μεν αντικείμενο της συμφωνίας, αλλά όσο σαφέστεροι είναι οι κανόνε ε, του παιχνιδιού είτε στην Κίνα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κινεζικέ επιχειρήσει, τόσο καλύτερο είναι. Διότι εμεί δεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ε, ε, πρωτοβουλία για το δρόμο του μεταξύ, θέλουμε όμω να έχουμε σαφείς κανόνε παιχνιδιού για όλου. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη διαπραγμάτευση αυτή τη συμφωνία μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο την πρωτοβουλία αλλά και τι χώρε τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες ε, ε, έχουν ξένες κινέζικες επενδύσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν υπογράψει και μνημόνια συνεννόησης βάσει ε, της συμφωνίας αυτής, κάποιοι άλλοι όχι. Ε, το να είναι σαφείς οι κανόνες του παιχνιδιού και ισότιμη όρια ανταγωνισμού βεβαίως ε, θεωρώ ότι βοηθάει όλους και τους επενδυτές. Ο κύριος Σόλτς. Η ερώτηση για τον ενεργειακό χάρτη. Ρωτήσατε αν θα φύγουμε. Προς το παρόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταρρυθμίσουμε τη συμφωνία και ε, συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις μεταρρύθμισης καλή την πίστη για να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να γίνει συμβατή με ό,τι θεωρούμε ότι είναι μια σωστή συμφωνία επενδύσεων. Δεν είμαστε σε στάδιο αποχώρησης ακόμα. Ε, η Ιταλία, για παράδειγμα, αποχώρησε από τη συνθήκη του ενεργειακού χάρτη, αλλά εμείς προς το παρόν θέλουμε να το μεταρρυθμίσουμε και να τη βελτιώσουμε. Ναι, η ρήτρα των κεκτημένων δικαιωμάτων, η τελευταία ερώτηση ήταν ε, για μένα για το, από τον ε, πρόεδρο, από τον κύριο Λάγκε, και αφορά τις διμερείς ε, επενδυτικές συμφωνίες των κρατών μελών. Βάσει του κανονισμού θα πρέπει εμείς να αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2020, στις αρχές του 2020, να υποβάλουμε έκθεση. Προφανώς και σκοπεύουμε να το κάνουμε και το σκεπτικό είναι όχι μόνο να υποβάλουμε την έκθεσή μας βεβαίω, αλλά και να ε, καθορίσουμε τα πιθανά επόμενα βήματα. Και τη δεδειμένη ε, χρονική στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να πούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να δούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος επίτροπος. Τους επόμενους μήνες νομίζω θα ξεκαθαριστούν αυτά. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ε, ή να το πω αλλιώ, ο κανονισμό για τα κεκτημένα δικαιώματα είχε διάφορε πτυχέ. Ο, μία πτυχή ήταν οι νέες συμφωνίε επενδύσεων που θέλουν να διαπραγματευτούν οι ε, χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που μπορούν να το κάνουν, ε, ειδικά με χώρες που δεν έχουμε συμφωνία, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό έχει επιτευχθεί γιατί όλες οι νέε διμερεί συμφωνίε επενδύσεων ακολουθούν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τι γίνεται με τις παλιές συμφωνίες Και οι παλιέ συμφωνίε δεν έχουν υποχρέωση απλώς να διαγραφούν. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται και, και κανονισμός και κτημένων δικαιωμάτων. Έχουν προστατευτεί ουσιαστικά. Θέλουμε να τις αντικαταστήσουμε σταδιακά, αλλά είναι χιλιάδες. Πάνω από χίλιες. Θα χρειαστεί λοιπόν χρόνος πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει σταδιακά να αντικαταστήσει όλες αυτές τις διμερείς συμφωνίες με όλους αυτούς τους εταίρους και να έχει μια ε, νέα προσέγγιση. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν να περιμένουμε μέχρι το 2030. Κόλλιν, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις για την επίλυση ε, επενδυτικών διαφορών. Η πρώτη ερώτηση της κυρίας Ροντρίγκης Πινέρο αλλά και του κυρίου Κανές Περές για το χρονοδιάγραμμα και τις προσδοκίες που έχουμε. Νομίζω πως βρισκόμαστε σε ένα στάδιο της διαδικασίας όπου βλέπουμε χώρες να υποβάλουν ιδέες και προτάσεις. Υπάρχουν διμερείς συζητήσεις που γίνονται στο περιθώριο των συναντήσεων αυτών. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε μια συγκεκριμένη σαφή πρόταση η προσπάθεια που θα καταβληθεί τους ερχόμενους μήνες με τις συναντήσεις του Οκτωβρίου, του Ιανουαρίου και του Απριλίου ενδεχομένω. θα γίνουν και στο πλαίσιο της συνενέσης που προσπαθούμε να επιτύχουμε, αλλά και κάπως παρασκηνιακά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τελικό στόχο. Θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να δούμε ποιες είναι οι κοινέ βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε την ε, συνένεση. Και είναι δύσκολο να κάνω μια εκτίμηση σχετικά με το πόσος καιρός θα χρειαστεί. Ίσως τον Ιανουάριο ενδεχομένως θα έχουμε καταλήξει ή μπορεί και τον Απρίλιο. Αλλά μετά το 2020, ίσως το 2021, μπορώ να εκτιμήσω ότι θα έχουμε φτάσει στον στόχο. Βέβαια, τον Ιούλιο θα πρέπει να εγκριθεί αυτή η συμφωνία προτού εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει πολλή δουλειά ακόμα μέχρι να περάσει ο φάκελος αυτός ε, στον ε, ΟΗΕ και υπογραφεί και περάσει μετά πάλι, επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικύρωση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε δύο-τρία χρόνια ακόμα τεχνικών εργασιών. Η κυρία Πέρες ρώτησε επίσης για τη συνέπεια. Το σκεπτικό πίσω από το πολυμερές ε, επενδυτικό δικαστήριο είναι να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ε, περίπου 3.000 επενδυτικές συμφωνίες. Ο μηχανισμός ε, λοιπόν αυτός θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ε, συμφωνίες αυτές και να προσαρμοστεί στην καθεμία. Και επειδή θα είναι ένας οργανισμός που θα αποφασίζει, θα δώσει αυτό και συνέπεια. Επίσης, κάτω από μία συμφωνία υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, οπότε θα ωφελήσει και σε αυτό το τομέα. Θα ωφελήσει όμως όχι μόνο τις ε, διεθνείς ε, υποθέσεις αλλά και τις ε, εγχώριες. Ο κύριος Σόλτς έκανε μία ερώτηση για τις υποχρεώσεις των επενδυτών. Ο Κάρλος ήδη αναφέρθηκε στην διαδικασία που λαμβάνει χώρα στη Γενέβη αυτήν την περίοδο. Το σκεπτικό είναι να υπάρχει ανοιχτή δικαιοδοσία και οι χώρες να έχουν τη δυνατότητα κάτω από αυτές τις επενδυτικές συμφωνίες να ε, επιλύνουν τις επενδυτικές τους διαφορές σε αυτό το πολυμερές δικαστήριο. Οι διεθνεί τους υποχρεώσεις, λοιπόν θα συνδέονται με αυτές τις επενδυτικέ συμφωνίες. Θα υπάρχει ένας μηχανισμός, τον οποίο θα χρησιμοποιεί το Διεθνές Πολυμερές Δικαστήριο. Η ουσία όμως, των ε, συζητήσεων αφορά τα όσα είπε ο Κάρλος και πάει λίγο πιο πέρα από αυτό. Η κυρία Ροντρίγκης Πενέρο ρώτησε επίσης και για την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία συμμετέχει στην ομάδα εργασία, είναι μάλιστα αρκετά ενεργή. Όπως σας είπα, έχουμε 106 χώρες που συμμετέχουν ενεργά. Υπάρχει δηλαδή υψηλό επίπεδο Η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή εκφράζει κάποιες ανησυχίες για το μόνιμο χαρακτήρα της ε, δομής του δικαστηρίου αυτού. Ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα εκτελήσονται στις ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Ιαπωνία και εξελίσσονται τα πράγματα. Τέλος. Και αριθμό ρώτησε για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλωσορίσει την απόφαση του Δικαστηρίου 1.17 για την επίλυση διαφορών, δικαστική επίλυση διαφορών. Ε, διεξήχθη μία νομική ανάλυση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Είναι όμως πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται για αλλαγές έτσι ώστε να μπορούν οι χώρες να εγκρίνουν περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι οι φυστάμενες συμφωνίες θα αποτελέσουν πρόβλημα. Σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομολογία σε σχέση με παλαιότερες αποφάσεις, οι χώρες είναι ελεύθερες να νομοθετήσουν. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εμπόδιο σε αυτό για την πολιτική κατά της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι θα παραμένουμε σε επαφή για αυτά τα θέματα, γιατί η επενδυτική πολιτική είναι σημαντικό στοιχείο του όλου παιχνιδιού και στο επανειδήν και σύντομα. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα και τελευταίο για σήμερα το πρωί, η 13, είναι και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλούνται να παραμείνουν μόνο οι βουλευτές, οι βοηθοί τους, ε, ε, ε, οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων καθώς και η γραμματεία, η βοηθή των